Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, νομίζω καλά θα κάναμε να αρχίσουμε. Μπορεί να καταφτάσει και κανένα συνάδελφο, ελπίζουμε τουλάχιστον πάρα πολύ. Και καλωσορίζω θερμότατα όλους σα ε, για τη συνέχιση τη συνεδρίασή μας. Έχουμε δημόσια ακρόαση το απόγευμα και ανταλλαγή απόψε με θέμα ακαδημαϊκή μετεκπαίδευση και ε, εκπαίδευση εξ αποστάσεως ως στρατηγική ε, για τη διαβίου εκπαίδευση και μάθηση. Είναι ένα θέμα αυτό που έχει πολλές πτυχές με το οποίο θα ασχοληθούμε και αφιερώνουμε πολύ χρόνο στις εργασίες μας. Εδώ μιλούμε για παιδεία ε, και εκπαίδευση κάθε είδους και κάθε τύπου. Και αυτό που μας ενδιαφέρει σήμερα είναι η μετακπαίδευση, η διαβίου μάθηση και η αποστάσεως ε, εκπαίδευση. Ως ε, συντονιστές αποφασίσαμε να κάνουμε μια έκθεση πρωτοβουλίας με εισηγητή τον κύριο Σφέρ, στον οποίο θα δώσω το λόγο πρώτον μετά τους ε, πυρογνώμονές μας. Γιατί είναι και η πρώτη ανταλλαγή απόψεων η ακρόαση αυτή για την έκθεση πρωτοβουλίας του κυρίου Σφέρ τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα μάλλον της σημερινής δημόσιας ακρόσης θα αντανακλώνται και στην έκθεση αυτή πρωτοβουλίας. Και είμαι βέβαιο ότι και ο κύριος Φέρ και οι σκιώδες ε, εισηγητές ε, θα τεντώσουν τα αυτιά τους σήμερα έτσι ώστε να σημειώσουν ε, τις προτάσεις και τις ιδέες που θα ακούσουμε στην σημερινή ακρόαση και ελπίζω σχετικά σύντομα να καταλήξουμε σε μια καλή έκθεση εδώ στην Επιτροπή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια. Χωρίς περαιτέρω λοιπόν καθυστέρηση θα ήθελα να σας συστήσω τους τέσσερις προσκεκλημένους μας. Έχουμε τον κύριο Χέλμοντ Χόιερ, πρώην πρίτανη ε, του ε, Πανεπιστημίου Εξαποστάσεως διαλογραφία ε, του Χάγκεν της Γερμανίας και θα μας πει πώς η ψηφιοποίηση θα διαμορφώσει και θα ασφραγίσει το μέλλον. Έχουμε στη συνέχεια τον κύριο Κέβιν Χέδρινγκτον που θα μιλήσει για τη διαβιδίου εκπαίδευση και το ρόλο ε, της ε, μάθησης αυτής ε, στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Στη συνέχεια έχουμε την κυρία Μάρκοτ Κλίνκνερ ε, από ένα πανεπιστήμιο που διδάσκει διαλογραφίες και εξαποστάσεως και θα μας μιλήσει για στρατηγικές ε, απαντήσεις σε δημογραφικές και άλλες αλλαγές. Και τελευταίος, χωρίς να είναι λιγότερο σημαντικός, είναι ο κύριος Τζορτζ Ούμπαχτ από ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων που διδάσκουν πάλι παρέχουν προγράμματα σπουδών εξαποστάσεως για να μας πει πώς μπορεί να γίνει αυτό στο διαδίκτυο, ποιο είναι το νομοθετικό πλαίσιο και το ρυθμιστικό πλαίσιο και μπορεί να μας δώσει και ιδέες για το τι μπορούμε να κάνουμε από πλευράς νομοθετικής και ρυθμιστικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ όλους θερμότατα που βρήκατε το δρόμο προς τη Βρυξέλλες σήμερα. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε μαζί σας την πραγματογνωμοσύνη σας και τις γνώσεις σας ειδικέ για το θέμα αυτό. Θα δώσω πρώτα το λόγο ε, στον κύριο Χόια. Παρακαλώ έκαστος 10 με 15 λεπτά το πολύ. Κύριε Χόιερ, έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, στην οποία ανταποκρίθηκα με χαρά. Ε, σε τούτη εδώ την ομιγύρη δεν θα πρέπει να συζητήσουμε για τη διαβίου μάθηση. Ε, γνωρίζουμε ότι ε, ένας στους δύο πολίτες δεν τελειώνει τον εργασιακό του βίο στο ίδιο επάγγελμα το οποίο ξεκίνησε. Άρα η ερώτηση είναι τι γίνεται με τα προσόντα, με τη μετακπαίδευση και η απάντηση είναι διαβίου μάθηση. Ωστόσο, ε, ευθύ εξ αρχή θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση ε, δύο πραγμάτων που συνδέονται στον τίτλο της ομιλίας μου. Διότι από τη μια πρόκειται ε, για την ακαδημαϊκή μετακπαίδευση ή την μετεκπαίδευση σε πανεπιστήμια και την εξαποστάσεως, παλιά λεγόταν διαλογραφία σε αυτή η εκπαίδευση. Δηλαδή, στο πανεπιστήμιο, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, περιγράφουμε ε, ένα πρόγραμμα σπουδών, ε, τριτοβάθμια εκπαίδευση με διπλώματα, με πτυχία. Ε, έχει συγκεκριμένες ομάδες στόχους αυτή για μεταπτυχιακά και αυτό αφορά κυρίως επαγγελματίες αλλά και εκείνοι που σπουδάζουν, φοιτητές, ε, είναι μεταπτυχιακοί, έχουν κατά κανόνα ένα πρώτο πτυχίο στην πανεπιστημιακή μετακπαίδευση. Τέτοιες προσφορές υπάρχουν ε, μονάδες διδακτικές ε, που δίνουν ένα πτυχίο και τελικά μάστερ ή και διδακτορικά. Αν δούμε τώρα τι γίνεται ε, με την, ε, τις σπουδές εξ Αυτό είναι η μέθοδος ε, διδασκαλίας και εκμάθησης. Δεν είναι το περιεχόμενο, δεν είναι το πρόγραμμα σπουδών όταν σπουδάζεις εξ αποστάσεως, ούτε το πρόγραμμα σπουδών και πώς αυτό εντάσσεται. Οι εξ αποστάσεως σπουδές έχουν και πάλι ομάδες στόχους, είναι κυρίως εργαζόμενοι, επαγγελματίες, αλλά όλο και περισσότερο άνδρες και γυναίκες ε, στην οικογένεια ή σε ειδικέ ε, συνθήκες. Ε, έχουμε τέτοιες δυνατότητες εξ αποστάσεως μάθησης και διδασκαλίας από το σχολείο μέχρι το πανεπιστήμιο και το μεταπτυχιακό. Και αυτό το πρόγραμμα διακρίνεται περισσότερο από τη μέθοδο και η διαφορά και λιγότερο από το περιεχόμενο. Συμπέρασμα όταν μιλάμε για ακαδημαϊκή μετακπαίδευση, αυτή ε, η πανεπιστημιακή μπορεί να είναι η συμβατική ε, στο αφιθέατρο ή εξ αποστάσεως, face to face. Ε, η εξ αποστάσεως είναι μια μέθοδος εκμάθησης και διδασκαλίας ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Και η προσφορά έχει να κάνει με διδακτικές μονάδες, με μαθήματα, Υπάρχουν ε, ανοιχτά πανεπιστήμια, όπως το πανεπιστήμιο το δικό μας στο Χάγεν, με μπάτσελορ, με μάστερ και αντίστοιχα πτυχία και μετακπαίδευση και μεταπτυχιακά, πάντα εξ αποστάσεως. Δηλαδή, σε όλες αυτές τις συζητήσεις θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ξεχωριστά αυτά τα δύο. Την εκπαίδευση που γίνεται μετά το πτυχίο στο ίδιο το πανεπιστήμιο και την εξ αποστάσεως. Η πανεπιστημιακή μετακπαίδευση είναι αναπόσπαστο ε, στοιχείο της διαβίου μάθησης. Οι εξαποστάσεως ε, σπουδές είναι ένα ε, σύγχρονο σύστημα σπουδών φοιτησής που ανταποκρίνεται στην κινητικότητα των φοιτητών σήμερα και επίσης προσφέρεται πάρα πολύ για τη διαβίου μάθηση για ανθρώπους που εργάζονται. Και τα δύο αυτά λοιπόν και στο Πανεπιστήμιο αλλά και εξ Ε, είναι κάποια συστήματα σπουδών που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και προσφέρουν και ισότητα ευκαιριών. Αυτό ήταν η διαφορά που έχουν τα δύο συστήματα. Τι κοινό έχουν τώρα. Η ψηφιοποίηση αφορά το μέλλον και της πανεπιστημιακής κλασικής εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, αλλά και της εξαποστάσεως. Αυτό πραγματικά θα σφραγίσει ε, το μέλλον. Είναι κλειδί η ψηφιοποίηση για την ε, μεταξέλιξη αυτών των ε, δύο τρόπων σπουδών. Και στο πανεπιστήμιο και στην εξαποστάσεως φοιτηση οι φοιτητές είναι κυρίως ενήλικες. Έχουν Κάποιου περιορισμούς και μεγάλους λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας, οικογένειας ή κοινωνική ζωή ευρύτερα. Και εδώ η ψηφιοποίηση ε, βοηθάει και τις δύο ε, δυνατότητες. Πάντα κάνω αυτή τη διάκριση, είτε είσαι στο πανεπιστήμιο είτε εξ αποστάσεων ε, ε, φυτάς, έχεις ε, πλέον από την ψηφιοποίηση. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία, μεγαλύτερη διάδραση Υπάρχουν διάφορα σενάρια ας πούμε, εκπάθησης που υποστηρίζονται από το διαδίκτυο. Αυτό έχει να κάνει και με το περιεχόμενο, έχει να κάνει και με την επικοινωνία και με τη δυνατότητα συνεργασίας των φοιτητών μεταξύ τους, των μεταπτυχιακών κλπ. Στην εξαποστάσεως ε, φίτηση ε, υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα όπως είπαμε ε, και είναι κάτι που επιτάσσει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Στο Πανεπιστήμιο στην ακαδημαϊκή φοιτήση συνδέεται καλύτερα βάλει με την ψηφιοποίηση ο κόσμος της εργασίας με το πανεπιστήμιο. Ε, δεν είναι στεγανά αυτά. Και με την ψηφιοποίηση μπορούμε να φτάσουμε και σε νέες ομάδες στόχους που μέχρι σήμερα ε, ήταν εκτός. Αυτό ισχύει και για τους δύο τρόπους, και για την εξαποστάσεω και για την ε, εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο και σε πολλές περιπτώσεις ε, είναι πραγματικά ευρύτερε οι ομάδε με την ε, ψηφιοποίηση και μεγαλύτερο ο αριθμό των φοιτητών. Παρ' όλα αυτά ε, υπάρχει δυνατότητα με την ψηφιοποίηση εξατομίκευση και ειδική προσοχή για κάθε φοιτητή. Γιατί έρχονται οι φοιτητέ και έχουν διαφορετική προέλευση, διαφορετική μόρφωση, μορφωτικό επίπεδο και διαφορετικό στόχο μορφωτικό όταν έρχονται στο πανεπιστήμιο. Και θα πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτό με επιστοποιητικά, με πτυχία, με διπλώματα ε, που μπορεί να είναι ένα πιστοποιητικό ή ένα μάστερ χωρίς να συνιστά αυτό τίτλο πανεπιστημιακό πτυχίο δηλαδή. Και επιπλέον η ψηφιοποίηση ε, ανοίγει δρόμους για άλλους πόρους, όπως είναι η ανοιχτή εκπαίδευση, open education ή κάποιες επιγραμμικές ε, σπουδές ε, που μπορούν να χρησιμοποιούν οι φοιτώντες. Για να αξιοποιήσουμε όμως όλο αυτό το δυναμικό της ψηφιοποίησης στην εκπαίδευση, χρειάζεται παροχή υπηρεσιών και παρακολούθηση και πλαισίωση των φοιτητών. Student services λέγεται αυτό. Δηλαδή δεν βγάζει ένα πρόγραμμα σπουδών στο διαδίκτυο για να σπουδάσει μόνο του ο Πάντα υπάρχει ένα άνθρωπο με τον οποίο είναι σε επαφή και ο οποίο ασχολείται μαζί του. Και στο μέλλον δηλαδή στα προγράμματα σπουδών και στι προσφορέ, ε, θα πρέπει ο καθένα ε, να ε, μιλάει για τι δεξιότητε που έχει σε θέματα επικοινωνία και media. Αυτό ξεκινά από το σχολείο ήδη σήμερα και θα πρέπει να ενταχθεί και στις παιδαγωγικές ακαδημίες και να εκπαιδεύονται και οι δάσκαλοι σε αυτό. Είναι οι πρώτοι λεγόμενοι πολλαπλασιαστές που δημιουργούν ε, τις ευκαιρίες για να αξιοποιήσουμε το δυναμικό στη συνέχεια. Όμως, για να το αξιοποιήσουμε πλήρως και να το εκμεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό, ε, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την παιδαγωγική, ε, με τη διδασκαλία και την πληροφορική. Χρειαζόμαστε ένα ε, νομικό πλαίσιο πανευρωπαϊκό, σαφές και συγκεκριμένο. Τι σημαίνει αυτό. Και για τους ε, διδάσκοντες και για τους φοιτητές θα πρέπει να υπάρχει ασφάλεια δικαίου σε σχέση με τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα, σε σχέση με δικαιώματα χρήσης, σε σχέση με ασφάλεια των δεδομένων και προστασία αυτών. αλλά να υπάρχει και απρόσκοπτη πρόσβαση σε κάποια στοιχεία χωρίς ε, μόρφη και φραγμός. Αυτά θα πρέπει να ρυθμίζονται νομικά, νομοθετικά, έτσι προστατεύεται και το διδακτικό προσωπικό και ε, ε, σπουδαστές. Και οι δύο αυτοί κλάδοι που σας ανέφερα ε, οδηγούν ε, σε κάποιες σπουδέ. σε ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών. Και θα πρέπει τα πανεπιστήμια στη συνέχεια να τα γνωρίζουν αυτά. Δηλαδή χρειάζεται ε, πρότυπο και προδιαγραφή και η αναγνώριση των πτυχίων. Από τις διδακτικές μονάδες, από τα πτυχία, από τα πιστοποιητικά Υπάρχει μια σύμβαση της Λισαβόνας, αλλά δεν αρκεί αυτή. Όλο και περισσότερο. Υπάρχουν και μεγάλες εταιρείες που όλο και περισσότερο ε, ε, μπαίνουν σε αυτά τα χωράφια και κάνουν δικές τους ε, προσφορές και εκπαίδευση. Και θα πρέπει εμείς να καταλάβουμε ότι έρχονται σε εμά φοιτητέ με κάποια προσόντα και με κάποια πτυχία και πιστοποιητικά που έχουν λάβει εκτός πανεπιστημίου. Αυτό επίσης θα πρέπει να ισχύει για την προσμέτρηση και για τον υπολογισμό δεξιοτήτων και προσόντων. Υπάρχει επίσημη εκπαίδευση, υπάρχει και ανεπίσημη. Ας πούμε, σα είπα, εκτό πανεπιστημίου κάποιος ε, έχει κάποια προσόντα που έχει αποκτήσει σε μια ανεπίσημη οδό που μπορεί να είναι στην ιδιωτική οικονομία εταιρεία. Θα πρέπει να ασχοληθεί ο νομοθέτης με αυτά τα θέματα γιατί τι θα γίνει αν στο μέλλον έχουμε κάποια πτυχία, πιστοποιητικά και διπλώματα και γνώσεις που έχει αποκομίσει κάποιος εκτός πανεπιστημίου. Και μπορεί κάποια μέρα η επαγγελματική ζωή αυτά να τα αξιολογεί υψηλότερα και να, και να τα ε, εκτιμά περισσότερο από ότι τα επίσημα πτυχία. Βλέπε Google University. Γι' αυτό χρειάζονται ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ευρωπαϊκές οδηγίες και κατευθυντήριες γραμμές για να μπορούν και τα πανεπιστήμια να ανταποκρίνονται τα επίσημα. Για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα δεν χρειάζεται μόνο να κάνουν προσπάθειες τα πανεπιστήμια τα ίδια, αλλά ε, φέρει ευθύνη και η ευρωπαϊκή πολιτική να επιτρέψουν στα πανεπιστήμια να απαντήσουν σε τέτοιου είδου προκλήσεις. Και κατά τη γνώμη μου, και τελειώνω με αυτό, με την τελευταία μου διαφάνεια, θα πρέπει να ασχοληθούμε με την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Να τα λαμβάνουμε υπόψη ε, στη στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαβίου μάθηση. Εγκαίρως να ξέρουμε ποιο είναι το σκηνικό, πώς διαμορφώνεται και πώς θα το θα αντιμετωπίσουμε και θα το πλησιάσουμε εμείς. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χόρε. Πάρα πολύ εντυπωσιακή η παρουσίαση αυτή που δείχνει ότι έχουμε ακόμα προκλήσεις πέρα από την παιδεία και την εκπαίδευση που πρέπει να συνυπολογίζουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τώρα θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Χέδερινγκτον για να μας μιλήσει και να μας κάνει τη δική του παρουσίαση. Ε, er Χρειάζεται αυτό το μαραφέτη για τις διαφάνειες. Ευχαριστώ πολύ. Θα σας μιλήσω για τη διαβίου μάθηση εκπροσωπώντας το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Εργάζομαι στο πανεπιστήμιο αυτό και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για το πώς λειτουργούμε και πώς προσεγγίζουμε την διαβίου μάθηση στο πανεπιστήμιο αυτό. Στη συνέχεια θα αναφερθώ στην σημασία που δίνουμε σε κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με την απασχολησιμότητα. Και θα δείτε πώς αντιμετωπίζουμε εμεί στο ανοιχτό πανεπιστήμιο αυτά τα ζητήματα. Λοιπόν, ως πανεπιστήμιο το οποίο ιδρύθηκε το 1969 έχουμε μια συγκεκριμένη αποστολή να είμαστε ανοιχτοί σε όσο δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, γεωγραφικούς χώρους, ιδέες και δημιουργήσαμε ένα νέο μοντέλο ένα νέο μοντέλο ανώτατης εκπαίδευσης του Νομένου Βασίλειο. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ανοιχτού πανεπιστημίου είναι ότι για τα προπτυχιακά μας προγράμματα δεν απαιτούμε συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισαγωγής. Οποιοςδήποτε μπορεί να εγγραφεί. Είμαστε το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε 175.000 φοιτητές το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. Διδάσκουμε σε φοιτητέ όχι μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά παντού στην Ευρώπη και παντού στον κόσμο. Δύο εκατομμύρια συνολικά φοιτητέ έχουν σπουδάσει σε εμά από το 1969, όταν ιδρυθήκαμε δηλαδή. Και το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 δώσαμε 15.000 πτυχία. Στα πλαίσια του Ηνωμένου Βασιλείου τώρα, οι σπουδαστές μερικής φοιτησής αντιστοιχούν στο 38% των στολικών φοιτητών. Μειώνεται βέβαια το ποσοστό αυτό και αυτό έχει να κάνει με το ότι αυξάνονται τα δίδακτρα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ξέρετε ότι υπήρξε πρόσφατη κυβερνητική απόφαση που αύξησε το ποσό των διδάκτρων. Έχουμε 4.000 ακαδημαϊκό προσωπικό, ερευνητικό, υποστηρικτικό προσωπικό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και περιλαμβάνονται βέβαια και οι ερευνητέ φοιτητέ, οι οποίοι ε, παρακολουθούν τη δουλειά των ε, εγγεγραμμένων φοιτητών. Απασχολούμε επίση 5.000 συνεργαζόμενου καθηγητέ, οι οποίοι παρέχουν διδασκαλία, καθώ επίση και οργανώνουν εξετάσεις και υποστηρίζουν βέβαια τους φοιτητές κατά τη φοιτησή τους. Προωθούμε τις προτεραιότητε της Βρετανικής κυβέρνησης για την διαβίου μάθηση. Επίσης ε, συμμετέχουμε σε συγκεκριμένα προγράμματα του ΕΒ Βασιλείου όσον αφορά την παροχή διπλωμάτων μέσω προγραμμάτων μαθητείας και μας απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της απασχολησιμότητας. Όπως σας είπα, ανέκαθεν είχαμε μια πολύ ανοιχτή πολιτική όσον αφορά την εγγραφή των φοιτητών και προσπαθούμε να προωθήσουμε μέσω των προγραμμάτων μας αυτών την κοινωνική κινητικότητα. Έχουμε ένα νέο στρατηγικό όραμα Προκειμένου να τα πετύχουμε όλα αυτά, θέλουμε να απευθυνθούμε όσο το δυνατόν περισσότερου φοιτητέ μέσω προγραμμάτων εκμάθηση που θα αλλάξουν πραγματικά τη ζωή του και που θα του βοηθήσουν να αποκριθούν στι ανάγκε του και να εμπλουτίσουν κατά αυτόν τον τρόπο την κοινωνία. Ποιο είναι το προφίλ των φοιτητών μα τώρα. Όπως σας είπα πριν από λίγο, έχουμε 175.000 φοιτητές αυτό το ακαδημαϊκό έτος. Το 77% των ανθρώπων αυτών δεν έχουν κάποια προσόντα νότα της εκπαίδευσης. Ουσιαστικά έρχονται στο ανοιχτό πανεπιστήμιο από πολλά διαφορετικά ακαδημαϊκά και κοινωνικά υπόβαθρα. Έχουμε φοιτητές από 18 μέχρι 90 ε, ετών. Η μέση ηλικία δεν είναι 29 έτη και η μέση αυτή ηλικία μειώνεται προϊόντος του χρόνου. Ένα 11% των φοιτητών μας προέρχονται από εθνοτικές μειονότητες, ενώ ένα 10% των φοιτητών μας έχουν δηλώσει ότι έχουν μια κάποια αναπηρία σωματική ή διανοητική. Και όσον αφορά το ζήτημα της απασχολησιμότητας, πάνω από το 75% φοιτητών μας εργάζονται σε καθεστώς πλήρους ημερικής απασχόλησης, ενώ φοιτούν σε εμά στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Με άλλα λόγια, διδάσκουμε πολύ συχνά σε φοιτητέ οι οποίοι ήδη εργάζονται. Το υπόλοιπο 25% είναι είτε φοιτητέ οι οποίοι είναι άνεργοι, είτε φοιτητέ οι οποίοι ασχολούνται με τη φροντίδα μελών της οικογένειας ή ηλικιωμένων μελών της κοινωνίας ή είναι συνταξιούχοι. Ποιο είναι τώρα το πρότυπο διδασκαλία το οποίο ακολουθούμε. Έχουμε ένα μείγμα μεθόδων διδασκαλία. Χρησιμοποιούμε επιγραμμικό, διδακτικό και έντυπο υλικό και χρησιμοποιούμε επίση παράδοση επιγραμμικών αλλά και διαπροσωπικών μαθημάτων ο φοιτητή δηλαδή μπορεί να βρίσκεται σε μια αίθουσα με τον καθηγητή να συνομιλεί με τον καθηγητή μέσω ιστοσελίδα. Έχουμε επιγραμμικά φόρουμ μέσω των οποίων μπορούν να έρθουν σε επαφή μεταξύ του οι φοιτητέ. Και επίση παρέχουμε και εκπαιδευτικέ ημερίδε ή μαθήματα τα οποία παραδίδονται σε εγκαταστάσει μα. Επίσης έχουμε εκπαιδευτικά μοντέλα και μοντέλα φίτηση τα οποία είναι ιδιαίτερα ευέλικτα. Δίνουμε τη δυνατότητα στου φοιτητέ να διακόπτουν τι σπουδέ του για ένα χρονικό διάστημα, να κάνουν κάποιο διάλειμμα αν αυτό απαιτείται και να επανέρχονται πάλι σε εμά. Και παρέχουμε επίση και ευέλικτε μεθόδου αξιολόγηση. Ουσιαστικά προσπαθούμε να έχουμε πάλι εδώ πέρα επιγραμμικά τεστ, επιγραμμικέ εξετάσει ή ακόμα και παράδοση εργασιών και συγκεκριμένων projects. Όπω σα είπα, είναι εντελώ ευέλικτο και ανοιχτό το σύστημά μας όσον αφορά την ε, ένταξη των φοιτητών στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Δεχόμαστε φοιτητέ ε, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν κάποια προπτυχιακά προσόντα. Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιου φοιτητέ ε, να συμμετέχουν σε αυτό το οποίο ονομάζουμε access courses, κάποια δείγματα, αν θέλετε, μαθημάτων, διδακτικών μονάδων, προκειμένου να δουν οι φοιτητέ αν όντω θέλουν να εγγραφούν. Προβλέπουμε συγκεκριμένα προγράμματα όσον αφορά του φοιτητέ με αναπηρίε και αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε ε, νέα προγράμματα προκειμένου να μειωθεί η υποεκπροσώπηση μαύρων φοιτητών ή εθνοτικών μειονοτήτων. Όσον αφορά την υποστήριξη τώρα των φοιτητών, πέρα από του καθηγητέ που βοηθούν του φοιτητέ, έχουμε και ερευνητέ φοιτητέ ή άλλου φοιτητέ ή καθηγητέ που προσπαθούν με διαδραστικό τρόπο να βοηθήσουν του φοιτητέ μα και προσπαθούμε επίση μέσω συστημάτων ανάλυση τη διαδικασία εκμάθηση να εντοπίσουμε τις πραγματικές ανάγκες των φοιτητών και να αναλάβουμε προφραστική ε, δράση προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά τους. Όπως και οποιοδήποτε άλλο πανεπιστήμιο στον Ηνωμένο Βασίλειο, έτσι και εμείς ε, υπαγόμαστε σε προγράμματα εξωτερικής αξιολόγησης ποιότητος, όπως άλλωστε προβλέπεται από τη Βρετανική νομοθεσία. Υπάρχουν εξωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι έρχονται και μας επισκέπτονται ανατακτικά χρονικά διαστήματα, όπως γίνεται και με τα κλασικά παραδοσιακά πανεπιστήμια και προφανώς προσπαθούμε και εμείς να προσαρμοστούμε με τις απαιτήσει του Βρετανικού κώδικα ποιότητος όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση. Όσον αφορά τώρα τη βελτίωση και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, χρησιμοποιούμε εμείς έναν ορισμό. Αναφερόμαστε σε ένα σύνολο ικανοτήτων και επιτευγμάτων που βοηθούν τους φοιτητές στη διαμόρφωση της σταδιοδρομίας τους, αυξάνοντας τις προσδοκίες τους και ενισχύοντας τη συμβολή τους στην κοινωνία. Όπως είπε και προλαλή σας, συνειδητοποιούμε και εμείς ότι όλο και περισσότερο οι πολίτες χρειάζεται να φοιτούν καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, ότι καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους θα έχουν πολλές διαφορετικές σταδιοδρομίες και ότι προφανώς η εργασία που είχαν όταν πρωτομπήκανε στην αγορά εργασίας δεν θα είναι η ίδια όταν θα φτάσουν στην ηλικία συνταξιοδότησης. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συμπληρωματική ακαδημαϊκή εκπαίδευση και εξαποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει πραγματικά τους φοιτητές όχι μόνο αυτούς οι οποίοι δεν κατάφεραν να πάρουν ένα πτυχίο στην ηλικία των 18 ή να αποφοιτήσουν από κάποιο λύκειο, αλλά και όλους τους υπόλοιπους πολίτες που θέλουν να αυξήσουν τις δεξιότητές τους. Ένα 85% των αποφύτων μας έχει δηλώσει ότι η φίτηση στο ανοιχτό πανεπιστήμιο τους βοήθησε πραγματικά να πετύχουν τους στόχους στα δεδρομία τους. Δεν λαμβάνουν λοιπόν μόνο θεωρητική εκπαίδευση αλλά και τις πραγματικές δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να εξελιχθούν επαγγελματικά. Γνωρίζουμε ότι έχουμε όλο και περισσότερους φοιτητές οι οποίοι θέλουν να σπουδάζουν μεταποδοχών, αν θέλετε. Ένα 76% των φοιτητών μας, όπως σας είπα, εργάζονται σε καθεστώς πλήρους ημερικής απασχόλησης. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το δικό μας το μοντέλο είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για τους ανθρώπους αυτούς που δεν θέλουν να αφήσουν τη δουλειά τους, να πάρουν άδεια άνευ αποδοχών προκειμένου να πάρουν κάποιο πτυχίο, να κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές. Και αυτό βέβαια βολεύει ιδιαίτερα τους ανθρώπους αυτούς που έχουν εξαρτώμενα μέλη και οικογένειες και 88 από τις 100 εισηγμένες στον δίκτυ Φούτσι εταιρείε έχουν ε, ενισχύσει οικονομικά το προσωπικό τους προκειμένου να μπορεί να φυτά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο ή να επιλέγει συγκεκριμένες διδακτικές μονάδες. Έχουμε τώρα και κάποιους ε, τομείς όπου προσπαθούμε να επικεντρωθούμε λίγο περισσότερο όσον αφορά το ζήτημα της απασχολησιμότητας. Έχουμε προγράμματα μαθητείας όσον αφορά τους ή τις νοσοκόμους ή συγκεκριμένα ε, προγράμματα κατάρτισης όσον αφορά την κοινωνική εργασία. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή το Ηνωμένο Βασίλειο προβλέπει ότι υπάρχουν ε, συγκεκριμένα προγράμματα χρηματοδότησης προκειμένου να δίδονται κίνητρα σε επιχειρήσεις να δέχονται ασκούμενους φοιτητές στα πλαίσια τους για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Εμείς συμμετέχουμε από τη δική μας πλευρά στα προγράμματα αυτά, προσπαθώντας να προωθήσουμε αυτά τα προγράμματα μαθητείας και κατάρτισης. Επίσης, σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών προσφέρουμε ένα MBA, Έχουμε δηλαδή προγράμματα επαγγελματική αδρομίας που επικεντρώνονται στη διαχείριση επιχειρήσεων και έχουμε επίσης και κάποιες διδακτικές μορφές οι οποίε είναι πιο άτυπε ή μη τυπικέ, αν θέλετε. Αναφέρθηκε σε αυτό και ο προηγούμενο ομιλητής. Παρέχουμε σύντομα προγράμματα εκμάθησης, ανοιχτά ή ανοιχτά μαζικά διαδικτυακά προγράμματα. Προσπαθούμε επίσης να εντάξουμε την συνιστόσα της απασχολησιμότητας σε όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Σε κάθε επίπεδο διδασκαλίας μας προσπαθούμε να έχουμε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων που θα επιτύχει, που θα αποκτήσει ο φοιτητή με την αποφύτιση από το πρόγραμμα αυτό. Κατά αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητέ μπορούν να διαμορφώσουν καλύτερα την επαγγελματική του ταδρομία, να αποκτήσουν συγκεκριμένε δεξιότητε, οι οποίε μάλιστα συμφωνούνται από κοινού με εργοδότε, οι οποίοι μα λένε ποιε είναι οι πραγματικέ του ανάγκε. Υπάρχει τώρα η Συνομοσπονδία Βρετανών Βιομηχάνων που έχει ε, καταρτήσει 7 συγκεκριμένες δεξιότητες που οι Βρετανοί βιομήχανοι θεωρούν ότι θα πρέπει να έχουν οι Βρετανοί πολίτες προκειμένου να, να βρουν πιο εύκολα μια θέση απασχόλησης. Αυτό που προσπαθήσαμε εμείς να κάνουμε είναι να πάρουμε τις 7 αυτές δεξιότητες και να τις ενσωματώσουμε στα προγράμματά μας, στα προγράμματα διδασκαλία μας. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι περισσότεροι φοιτητές μας θα καταφέρουν να αποκτήσουν αυτές τις δεξιότητες. Αυτά είναι τα ωφέλη τα οποία έχουμε εντοπίσει εμεί όσον αφορά την συμπληρωματική εκπαίδευση και την εξαποστάσεω εκπαίδευση, ιδίω όσον αφορά τον δείκτη τη αποσχολησιμότητα, Μπορούν να φοιτούν σε εμά οι ε, φοιτητέ μα ενώ παράλληλα εργάζονται δεν χρειάζεται λοιπόν να εγκαταλείψουν το χώρο εργασία του. Επίση, μπορούμε να ενισχύσουμε κατά αυτόν τον τρόπο την απασχολησιμότητα, δίνοντα τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερου ανθρώπου να συμμετέχουν στα προγράμματά μα, ανεξάρτητα από το κοινωνικό-οικονομικό του υπόβαθρο, ανεξάρτητα από τι αναπηρίε που ενδεχομένω να έχουν ή τι ευθύνε φύλαξη εξαρτωμένων μελών. Η επιλογή λοιπόν αυτή του ανοιχτού πανεπιστημίου είναι πολύ πιο φτηνή, πολύ λιγότερο δαπανηρή σε σχέση με τα κλασικά παραδοσιακά πανεπιστήμια. Προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο με καινοτόμο τρόπο τι νέε μορφέ τεχνολογία. Προσφέρουμε συγκεκριμένα προγράμματα, πολλέ φορέ προσαρμοσμένα στι ανάγκε των φοιτητών. Προωθούμε επίση ε, μαζικά ανοιχτά προγράμματα εκμάθηση. Προσπαθούμε επίσης να δώσουμε τη δυνατότητα στους φοιτητές μας να συνδυάσουν την εμπειρία που ενδεχομένω να έχουν ήδη αποκτήσει σε άλλους επαγγελματικού χώρους με τη δική μας θεωρητική εκπαίδευση στα πλαίσια του Πανεπιστημίου και προσπαθούμε κατά αυτόν τον τρόπο να προωθήσουμε τόσο τις επαγγελματικές και προσωπικές ανάγκες των φοιτητών μας αλλά και να ανταποκρίνονται αυτές τις ίδιες τις ανάγκες της κοινωνίας. Θα ήθελα ή δυνατόν τώρα να σας δείξω ένα σύντομο φιλμάκι που έχουμε γυρίσει όσον αφορά το ρόλο του ανοιχτού πανεπιστημίου.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 Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ εντυπωσιακά αυτά που ακούμε και μας δείχνει ουσιαστικά πώς λειτουργεί ένα τέτοιο ανοιχτό πανεπιστήμιο και πώς εγγράφεται στην πραγματική ζωή. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και πώς μπορεί κανείς να συνδυάσει ε, την επαγγελματική του ζωή με τη φίτηση στο ανοιχτό πανεπιστήμιο. Και τώρα με χαρά θα ακούσουμε την κυρία Κλίνκνερ, στην οποία δίνω αμέσω το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σα κυρίε και κύριοι. Καταρχά θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ στην ακρόαση αυτή και την ευκαιρία που μα δίνετε να ακούσετε τα μελήματά μα και τι θέσει μα. Λέγομαι Μάργκοτ Κλίνκνερ, εργάζομαι ε, στη ε, πόλη Koblenz ε, εκπροσωπώ τη γερμανική κοινωνία και εταιρεία για την μετεκπαίδευση και την ε, εξαποστάσεως φίτηση. Και ο πρόεδρος της εταιρείας, κύριος Μπορχατλίμαν με συνοδεύει σήμερα εδώ. Τέσσερα θέματα θέλω να σας αναφέρω και να σας εξηγήσω. Τι μας ενδιαφέρει. Να σας παρουσιάσω σύντομα το σύλλογο μου Γερμανικό σύλλογο ε, Πανεπιστημίων για την ε, Μετεκπαίδευση και την εξαποστάσεω Εκπαίδευση. Το δεύτερο είναι τα βασικά μας ε, στοιχεία και τι ζητάμε για μια στρατηγική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα συμπεράσματα. Η γερμανική εταιρεία λοιπόν ε, για την μετακπαίδευση και την εξαποστάσεως εκπαίδευση είναι ένα σύνολο που συγκεντρώνει πάνω από 300 ιδρύματα πανεπιστημιακά ανώτατης εκπαίδευσης στην ε, Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία. Εκπροσωπούμε ε, προγράμματα μεταπτυχιακά και μετακπαίδευσης επιστημονικής και για να μπορέσουμε να εγγραφούμε στο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία και να βοηθήσουμε χρησιμοποιούμε πολλά κανάλια, πολλούς, διά, πολλούς διάβλους ε, επικοινωνίας και συνεργαζόμαστε σε διάφορα επίπεδα με διαφόρους φορείς. Συγγνώμη κυρία Κλίνκνερ, αλλά εδώ μου ανάβει ένα φωτάκι γιατί τρέχετε. Θα πρέπει να μιλάτε λίγο πιο αργά γιατί δεν θα σας προλάβουν οι διερμηνείς μας. Ναι χρησιμοποιούμε διάφορους διάβλους επικοινωνίας και μορφοτύπους εργαζόμαστε ε, και συνεργαζόμαστε σε διάφορα επίπεδα με διάφορους ενδιαφερομένους και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή δομή που είναι ένα δίκτυο για την ε, διαβίου μάθηση. Τι γίνεται με την ψηφιοποίηση. Το ακούσαμε προηγουμένως και στις δύο τοποθετήσεις και για μας έχει ε, πολύ μεγάλη σημασία αυτό και εστιάζουμε στην προσπάθειά μας. Εμείς εκπροσωπούμε ε, τα πανεπιστήμια και συγκεκριμένα τη διαβίωμα μάθηση και τη μετακπαίδευση και είμαστε πεπισμένοι ότι η επιστημονική αυτή ε, εκπαίδευση θα πρέπει να απαντά στη δημογραφική αλλαγή και στην τεχνολογική αλλαγή της κοινωνίας μας. Αλλάζουν και τα επαγγέλματα και ο τρόπος εργασίας. Και είναι μεγάλη οι προκλήσεις να ε, σας ε, παρουσιάσω κάποια βασικά στοιχεία και αρχές μας. Η συμπληρωματική ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ACE, είναι εκπαίδευση που προσφέρουν τα πανεπιστήμια. Αυτό ε, αφορά επαγγελματικά προσόντα, αλλά και γενική ακαδημαϊκή εκπαίδευση. Ποιες είναι οι ομάδες στόχοι. Είναι πολύ ευρύ το φάσμα. Μπορεί να είναι πτυχιούχοι πανεπιστημίου ή μπορεί να είναι ε, άνθρωποι που έχουν επαγγελματική εμπειρία ή εργαζόμενοι που δεν έχουν φοιτήσει ποτέ σε πανεπιστήμιο. Ε, οι προσφορές επίσης αφορούν και κάποιους που έχουν εγκαταλείψει ε, κάποια στιγμή την εργασία τους για λόγους οικογενειακούς ή άλλους και επανέρχονται. Ή άνθρωποι που έχουν βγει στη σύνταξη και είναι ηλικιωμένοι ή αυτή τη στιγμή είναι και πρόσφυγες. Άρα η ε, ομάδα στόχη είναι πολύ διαφορετική, η προσφορά είναι πολύ διαφορετική και με την προσφορά μας βοηθούμε και ε, ε, στην ένταξη και στην καταπολέμηση του αποκλεισμού στην κοινωνία. Η επαγγελματική κατάρτιση και μετακπαίδευση στη Γερμανία και στην Ευρώπη βασικά δεν είναι κάτι που εμείς αντιλαμβανόμαστε ως συνέχεια της επαγγελματικής κατάρτισης, αλλά είναι και επιστημονική μετακπαίδευση ε, και είναι ένα είδος επαγγελματικού προσανατολισμού. Ε, τα αρχικά στα αγγλικά είναι HCVT. Ε, αυτό είναι η συνέχιση ε, της επαγγελματικής κατάρτισης που προτείνει το Πανεπιστήμιο και πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε ε, αυτό όταν μιλάμε για επαγγελματική κατάρτιση, ότι είναι μια μετακπαίδευση πανεπιστημιακού επίπεδου. Και πάλι έχουμε διάφορες ομάδες στις οποίες απευθυνόμαστε. Και είναι ένα τμήμα του ULLL που είναι η διαβίου μάθηση στο Πανεπιστήμιο. Στην ψηφιακή εποχή λοιπόν θα πρέπει συνειδητά να χρησιμοποιούμε ε, τις δυνατότητες που έχουμε για να είναι πιο ευέλικτοι ε, οι τρόποι διδασκαλίας και εκμάθησης. Τα είπε πολύ ωραίο ο κύριος Χόιερ και ο προλαλής σας. Ε, ακριβώς για να μπορεί κανείς να συνδυάζει το επάγγελμα, την οικογένεια και τις σπουδέ, ανεξαρτήτως ηλικίας και επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Στο στάδιο δηλαδή που βρίσκεται κάθε φορά έτσι μπορούν να ε, μετακπαιδεύονται, να μορφώνονται σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους οι εργαζόμενοι ή μη εργαζόμενοι. Ε, εκεί είναι η στρατηγική απάντηση. Και πάλι τρέχετε πάρα πολύ. Δεν σας προλαβαίνουν οι διερμήνες. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι επειδή βλέπω και το ρολόι. Yeah. Ähm, ich möchte auf Λοιπόν, τώρα θα ήθελα να επικεντρωθώ σε πέντε βασικές ε, αρχές, αιτήματα καλύτερα, ε, που θεωρούμε εμείς σημαντικά για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική της διαβίου μάθησης. Πρώτο σημείο. Επιστημονική μετεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση και μετεκπαίδευση είναι και διαφορετικά πράγματα, αλλά ε, ισότιμα. Το ανοιχτό πανεπιστήμιο από τη φύση του ε, βοηθάει να υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα και μεγαλύτερη ισότητα και ισότητα ευκαιριών ε, στην επαγγελματική ζωή. Κατά την άποψή μας, θα πρέπει να συνδέσουμε την επαγγελματική κατάρτιση ε, και την επιστημονική μετακπαίδευση καλύτερα. Δηλαδή, να μην διαχωρίζουμε πανεπιστήμιο και επαγγελματική κατάρτιση. Ίσα ίσα θα πρέπει ε, να υπάρχει αλληλοδιείσδυση αυτών των ε, συστημάτων. Πώς θα γίνει αυτό με αμοιβαία αναγνώριση των διαφόρων κλάδων και τομέων. Ότι είναι ισότιμη και εισάξιοι. Το ακούσαμε και προηγουμένως. Δηλαδή υπάρχουν και κάποιες άτυπες ε, μορφές μάθησης και διδασκαλίας και κάποια πιστοποιητικά που δεν είναι πτυχία. Άλλο θέμα που μας ενδιαφέρει μας είναι η επιστημονική μετεκπαίδευση είναι και παραμένει μη εμπορικού χαρακτήρα. Είναι ένα τμήμα του πανεπιστημίου, ε, είναι ένα τμήμα της δουλειάς του πανεπιστημίου, όπως η έρευνα ε, και όπως οι δημοσιεύσεις. Δηλαδή δεν είναι εμπορικού χαρακτήρα, δεν έχει σκοπό το κέρδος. Εμείς έχουμε λάβει ε, θέση σε σχέση με αυτό και ε, σε σχέση με τις κρατικές ενισχύσεις. Από την άλλη, στην επαγγελματική κατάρτιση υπάρχει μια διάκριση στη ε, μετακπαίδευση και στη συνεχιζόμενη εκπαίδευση να αποκτήσουν περισσότερα προσόντα και δεξιότητες ή πιο σύγχρονα. Άλλο αίτημά μας. Η χρηματοδότηση της διαβίου μάθησης στα πανεπιστήμια θα πρέπει να ενταχθεί στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με νέα ε, προγράμματα σπουδών, με ψηφιακό περιεχόμενο ε, για μεγαλύτερη πρόσβαση για να μπορεί κανείς να συνδυάζει καλύτερα την επαγγελματική ζωή, την οικογένεια και τις σπουδές. Και επειδή και η ε, επαγγελματική κατάρτιση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο και ε, για τα πανεπιστήμια. Έχουμε νέες αλλαγές, είπαμε, σε επίπεδο τεχνολογίας, σε επίπεδο δημογραφίας, άρα αποκτά μεγαλύτερη σημασία και η μετακπαίδευση στα πανεπιστήμια. Δεν είναι μόνο οι προπτυχιακές σπουδέ. Θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση και συστηματικά να ε, χρηματοδοτεί και να προωθεί ε, τις ε, δραστηριότητες αυτές. Τέταρτον. ποιοτικό έλεγχο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ενιαίε προδιαγραφέ. Το ακούσαμε και προηγουμένω. Στην εποχή τη ψηφιοποίηση, ε, ε, η διαδικασία αυτή είναι διασυνοριακή και γνωρίζουμε και το σύστημα με το σύστημα της Μπολόνια ε, βασικός και κοινό στόχος είναι ο ενιαίος εκπαιδευτικός χώρος. Άρα χρειάζονται νέες προδιαγραφές, νέα πρότυπα και αυτό απαιτεί περισσότερο από ποτέ ποιοτικό έλεγχο. Αυτό έχει σημασία για να αναγνωρίζονται κάποιοι τίτλοι που δίνονται ή πιστοποιητικά εκτός πανεπιστημίου. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ισχύει ακόμα. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την μετεκπαίδευση στο πανεπιστημίο είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στη Γερμανία αναγνωρίζεται περίπου το 50% των εξωπανεπιστημιακών ε, ε, τίτλων. Ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο αρκεί να έχει φωτίσει κανείς μέχρι 7 μήνες ένα πανεπιστήμιο για να πάρει τίτλο bachelor. Εφόσον έχει πιστοποιητικά εκτός πανεπιστημίου. Ένα πέμπτο και τελευταίο να ενταχθεί αυτή η μετακπαίδευση στα πανεπιστήμια στην στρατηγική ψηφιοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παιδεία και το πανεπιστήμιο αναγνώρισε πάρα πολύ νωρίς ότι ε, αυτός είναι ένας κλάδος και ένας τρόπος που ε, θα επιτρέψει στο μέλλον σε πολλούς πολίτες και πολύ περισσότερους ε, να έχουν πρόσβαση στο πανεπιστήμιο εξ αποστάσεων με μαζικά μαθήματα, μαζικές σπουδές και το Open Education. Μια στρατηγική λοιπόν ψηφιοποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριλαμβάνει και τη διαβίου μάθηση στα πανεπιστήμια, σε επιστημονικό επίπεδο. Τελειώνω και φτάνω στα συμπεράσματα και στην προοπτική και πάλι επαναλαμβάνω τα πέντε βασικά ε, σημεία για μας ε, η επαγγελματική κατάρτιση και η μετακπαίδευση σε επαγγελματικό και σε πανεπιστημιακό επίπεδο πρέπει να συνδέονται. Δεύτερον, θα πρέπει να είναι ένα τμήμα ε, της εντολής που έχουν διανόμουν τα πανεπιστήμια και η ε, Ε, θα πρέπει να χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να υπάρχει ποιοτικό έλεγχος με ε, ορόσημα και η διαβίω εκπαίδευση να ενταχθεί οπωσδήποτε στην στρατηγική ψηφιοποίηση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας κυρία Κλίνκνερ. Πολύ εντυπωσιακά αυτά που μας λέτε κι εσείς και ιδιαίτερα με τα αιτήματά σας που είναι σαφέστατα και ξεκάθαρα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, θα ακούσουμε τον τελευταίο μιλητή, τον κύριο Ούμπαχτς. Έχετε το λόγο. Καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκπροσωπώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Εξαποστάσεως Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 12 ανοιχτά πανεπιστήμια εκπροσωπούμε συνολικά στην Ευρώπη και 12 με 15 ενώσεις και συλλόγους. και συμβατικών πανεπιστημίων, όχι μόνο ανοιχτών πανεπιστημίων, που προσφέρουν εξ υπηρεσίες μαθήματα. Εάν έχω και τις διαφάνειες, θα σας δείξω σήμερα τα αποτελέσματα μιας μελέτης μεταξύ των μελών μας για την ε, ε πιστοποίηση και την ε, εξασφάλιση της ποιότητας ε, που κάναμε στα πλαίσια της μελέτης της Κομισιόν για το μεταβαλλόμενο παιδαγωγικό πεδίο. Σχετικά λοιπόν με μαθήματα που παρέχονται στο διαδίκτυο ή εξ αποστάσεως. Η εξασφάλιση της ποιότητας, η διασφάλιση της ποιότητας ε, για τους ε, διαφόρους οργανισμούς πιστοποίησης και φορείς πιστοποίησης που οδηγούν σε διάφορες συστάσεις που προκύπτουν από τη μελέτη αυτή. Κοιτώντας καταρχά τα εθνικά πλαίσια και τις εθνικές διατάξεις, βλέπει κανείς ότι είναι πολύ ανοιχτά τα εφισταμένα πλαίσια για τα εξαποστάσεως μαθήματα, την εξαποστάσεως φίτηση. Αναγνωρίζονται σχεδόν παντού αυτά τα μαθήματα. Από την άλλη μεριά όμως, μόνο το ίμιση των κρατών έχει συγκεκριμένες διατάξει για την εξαποστάσεως φίτηση. Το οποίο σημαίνει ότι στις χώρες που δεν έχουμε συγκεκριμένες διατάξεις δεν έχουμε και στρατηγικές ή κίνητρα για, μια, για ένα σύστημα πιο καινοτόμο εκπαιδευτικό που θα κινείται και προς την ως φίτηση. Δηλαδή θα μπορούσαν να, να υπάρχουν και διατάξεις που αποτρέπουν δημιουργία νέων μαθημάτων ή καθηγητών. Εάν υπάρχει δηλαδή απέτηση παρουσίας του σπουδαστή και του καθηγητή διαζώσης. Πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα παρέχουμε κίνητρα και δεν θα παρεμποδίζουμε πιο ευέλικτες μορφές εκπαίδευσης. Για την διασφάλιση ποιότητας εντός της μελέτης βλέπουμε ότι η πλειοψηφία επικεντρώνεται σε κλασικά μαθήματα ή στους χώρους των πανεπιστημίων. Υπάρχουν όμως και κριτήρια για ανάμεικτα συστήματα σπουδών και εξ και στους χώρους των πανεπιστημίων. Εμείς ερευνήσαμε λοιπόν ενδείξεις καλών πρακτικών σχετικά με ανάμεικτα προγράμματα σπουδών και, καθό, και κατά πόσον παρέχονται από τα πανεπιστημία ε, κατευθυντήριες γραμμές. Σε κάποιες χώρες, Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Κύπρο, υπάρχουν πράγματι κατευθυντήριες ε, γραμμές που παρέχονται από τους κρατικούς φορείς στα πανεπιστήμια σχετικά με καινοτόμα προγράμματα φίτησης και εξ φίτηση. Όταν οι φορεί διασφάλισης ποιότητα υπάρχει πάνελ ειδικών, εκεί συμπεριλαμβάνονται και εμπειρογνώμονες ε, εξωτερικοί αξιολογητές, το οποίο ε, είναι καθησυχαστικό Γιατί εμείς θεωρούμε ότι μέσα στις διατάξεις, μέσα στους κανονισμούς αυτούς θα πρέπει να υπάρχουν και ρήτρε που να διευκολύνουν ή να προαγάγουν τα καινοτόμα προγράμματα εξεποστάσεως ε, φίτησης. Τώρα, οι, οργαν... κρατικοί φορείς ε, διασφάλισης ποιότητας και οι άλλοι φορείς διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να εξασφαλίσουν ε, ότι θα υπάρχει ενεργό συμμετοχή ε, της καινοτομίας εντός των προγραμμάτων σπουδών. Θεωρούμε ότι και τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά δίκτυα που έχουμε στην Ευρώπη θα πρέπει να βοηθήσουν την προσπάθεια αυτή ώστε να υπάρχει μια ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και ώστε να καθοριστούν ορισμοί στο πεδίο αυτό. Να μην μιλούμε δηλαδή για αόριστα πράγματα επί τη βάση αόριστων ορισμών και αποκλήσεων μεταξύ των κρατών μελών. Και για να κάνουμε ένα βήμα ακόμα πρέπει να ε, αναπτύξουμε ένα σύστημα συγκριτικής αξιολόγησης, benchmarking για να το πούμε ελληνικά, ώστε να αναπτύξουμε νέες μορφές εκμάθησης. Γιατί οι διαφορετικές χώρες της Ευρώπης έχουν και διαφορετική πρόοδο στην ανάπτυξη αυτών των προγραμμάτων σπουδών. Και χρειάζεται περισσότερη και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των χωρών σε αυτό το επίπεδο. Εάν υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των μη παραδοσιακών αυτού του είδους σπουδαστών και φοιτητών ή των φοιτητών παρακολουθούν μαθήματα ειδικών ορών αυτοί, αυτού του είδους οι σπουδαστές έχουν διαφορετικές ανάγκες από τους ε, σπουδαστές που παρακολουθούν στα κλασικά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων. Χρειάζονται λοιπόν πιο ευέλικτα ωράρια μεταξύ άλλων. Και εδώ το, το είναι ότι οι οργανισμοί διασφάλισης ποιότητας προσπαθούν, έχουν εντός των κανονισμών τους ε, τις προβλέψεις ώστε να προσπαθούν να συμπεριλάβουν και αυτό το κριτήριο στην αξιολόγησή τους. Δηλαδή το κριτήριο της ευελιξίας. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ε, η πτυχή της συνεχούς ε, εξειδίκευσης και κατάρτισης του προσωπικού. Ώστε ε, να έχει καταρτιστεί και στις νέες ευέλικτες μορφές εφήτησης. Βεβαίως οι θεσμικές στρατηγικές είναι η ρακοκαλιά της ε, καινοτομίας. Έχουμε προχωρήσει σε πολλές μελέτες σε όλες τις χώρες και πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ δύσκολο να διατρέξει κανείς μια ολόκληρη οργάνωση σε διάφορα επίπεδα προσωπικού και προγραμμάτων και πανεπιστημιακών σχολών. Υπάρχουν άλλοι φορείς υπό την αιγίδα των οποίων ή εντός του δικτύου των οποίων θα μπορούσε να ολοκληρωθεί επιτυχώς μια τέτοια προσπάθεια. Σε αυτή τη ε, διαφάνεια βλέπουμε ότι οι οργανισμοί διασφάλισης ποιότητας θα πρέπει να εξετάζουν το πλαίσιο, το προϊόν που παρέχει αν θέλετε το πανεπιστήμιο και τις ανάγκες των φοιτητών. και τον καινοτόμο χαρακτήρα της κάθε, του κάθε πανεστημιακού φορέα. <clears throat> Για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας θα πρέπει να αναπτύξουμε καινοτόμες στρατηγικές για νέες μορφές φοιτησης. Συχνά τα πανεπιστήμια εντάσσουν δραστηριότητες ε, διαδικτύου εντός των χώρων των πανεπιστημίων αυτό όμως δεν είναι ιδιαίτερα καινο, ε, καινοτόμο, γιατί όταν μιλούμε για νέες ε, εναρκτικές ή ευέλικτες μορφές εφήτησης, μιλάμε για την βελτίωση και όχι την αντικατάσταση βεβαίως της ε, εκπαίδευσης. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη και το προσωπικό. Και βέβαια υπάρχει και η ίδια η διαδικασία της πιστοποίησης ή της έκδοσης του οποιοδήποτε τίτλου που θα πρέπει να γίνεται με τους ίδιους κανόνες όπως και με τα κλασικά προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων, αλλά με τη χρήση διαφορετικών δικτών και κριτηρίων που να είναι συγκεκριμένα για τα προγράμματα εξ αποστάσεως Και ως Ευρωπαϊκό Σύνδεσμος έχουμε αναλάβει και αυτό το καθήκον να αναπτύξουμε τι σημαίνει και πόσο καλό μπορεί να είναι ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως ε, φοιτησης. Έχουμε αναπτύξει λοιπόν δείκτες και συγκριτική αξιολόγηση που τους ε, παρέχουμε στους οργανισμούς ε, διασφάλισης ποιότητας. Το ονομάζουμε e-excellence. Είναι ένα μέσο λοιπόν συγκριτικής αξιολόγησης που έχουμε επικαιροποιήσει ήδη δύο φορές τρεις φορές τα τελευταία δέκα χρόνια. Είναι open source και προσπαθούμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε έναν άμεσο σύνδεσμο με τα πανεπιστήμια ώστε να τα καθοδηγήσουμε στην επόμενη φάση της καινοτομίας. Έχουμε πλέον 75 εμπειρογνώμονες που εργάζονται στις ομάδες αξιολόγησής μας και παρακολουθούν στενά τι συμβαίνει στο πεδίο και ε, συνεργάζονται στενά με καθένα από τα πανεπιστήμια με τα οποία συνεργαζόμαστε και είμαστε σε επαφή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας κύριε ε, Κουρμπάχ. Σας ευχαριστώ όλους και τους τέσσερις ε, που ακριβώς εστιάσατε στα αιτήματα. Τι περιμένετε από εμά, τι ζητάτε από εμά, τι προτείνετε να κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη, που δεν πρέπει να ανακαταυτεί η Ευρώπη, τι πρέπει να κάνουν τα κρατημέλη. Ε, πάρα πολύ γόνιμα όλα αυτά για μας και πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ και για την έκθεση πρωτοβουλίας. Και είμαι βέβαιη ότι κάποια στιγμή κάτι από αυτό που ακούσαμε θα το ξαναβρείτε και στην έκθεσή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Σφαία, τον εισηγητή μας, για να μας πει τις πρώτες σκέψεις του για την έκθεση πρωτοβουλίας, πώς σκέφτεται να την ε, καταρτήσει και να την εκπονήσει. Μετά θα ακούσουμε τους και ηγητέ και τους υπολείπους. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι καλεσμένοι μας, καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις εξαιρετικές αυτές παρουσιάσεις που μας κάνατε. Ειλικρινά σας λέω ότι έμαθα πολλά χρήσιμα πράγματα σήμερα το απόγευμα μας δώσετε πραγματικό μάθημα, θα έλεγα, στον τομέα αυτό που πρέπει και εμείς να δραστηριοποιηθούμε περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες, καθότι θέλουμε να καταρτήσουμε μία πολύ καλή έκθεση για αυτό το ζήτημα. Όσοι ασχολούνται με τον τομέα της παιδείας και της εκπαίδευσης προσπαθούν να πετύχουν δύο γενικούς στόχους. Πρώτον, βελτίωση της παρεχόμενης παιδείας, καλύτερη αποτελεσματικότητα και καλύτερη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό αυτό σύστημα σε όσο δυνατόν περισσότερους πολίτες. Ζούμε σε έναν κόσμο και σε μια κοινωνία που μεταβάλλεται συνεχώς. Απαιτείται πλέον να αναβαθμίσουμε συνεχώς τις ικανότητες και τις γνώσεις μας. Ακούσαμε ότι το πτυχίο το οποίο λάβαμε κατά τη διάρκεια των ανικών μας χρόνων, δεν αρκεί πλέον και ότι αποτελεί απλώς την εφετηρία για τη μετέπειτα εξέλιξή μας και ότι τελικά η όλη διαδικασία της εκμάθησης είναι μία αένεη διαδικασία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο και περισσότεροι πολίτε να μπορούν να ενταχθούν στα προγράμματα διαβίου μάθηση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και από οικονομική αλλά και από κοινωνική πλευρά. Ένα από τους καλεσμένους μας το είπε πριν από λίγο ότι ακόμα και η επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση απαιτεί πλέον να συνεχίζουμε να εκπαιδευόμαστε, να αναβαθμίζουμε τις επαγγελματικές μας γνώσεις, ιδίως αν θέλουμε να μπορούμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τις νέες αυτές αναδυόμενες τάσεις της ε, οικονομίας. Ο Ανδρέας Σλάιντερ από τον ΩΣΑ έγραψε πριν από λίγο και τον παραθέτω, ότι η επαγγελματική κατάρτιση έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Το να καταρτίζει και να εκπαιδεύει κανεί όμω κάποιον πολύ νωρί για να κάνει μόνο μία δουλειά για όλη τη ζωή του δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση απάντηση στι απαιτήσει τη διαβίου μάθηση. Ανταυτού, αυτό το που χρειαζόμαστε είναι καλύτερη διασύνδεση ανάμεσα στα προγράμματα εκπαίδευση και την αγορά εργασία. Θα πρέπει να υπάρχει μια ομαλή μετάβαση από το εκπαιδευτικό σύστημα στην αγορά εργασία. Αφενό, και αφετέρου θα πρέπει να ενισχύσουμε τους πολίτες προκειμένου να αποκτούν κατά τη διάρκεια της πνευματικής τους ζωής όλο και περισσότερες δεξιότητες. Η σημερινή μας λοιπόν δημόσια ακρόαση θα επικεντρωθεί επίσης και στον ρόλο που διαδραματίζει η εξαποστάσεως εκπαίδευση και η επιγραμμική διαδικτυακή εκπαίδευση αν προτιμάτε. Η εκπαιδευτική αυτή μέθοδος έχει πάρα πολλές νέες δυνατότητες. Πρόκειται για μια νέα μέθοδο απόκτησης γνώσεων, μια νέα μέθοδο διδασκαλίας και νομίζω ότι το δυναμικό εδώ πέρα είναι τεράστιο. Πρόσφατα πήγα σε ένα καταπληκτικό μάθημα που έδωσε η κυρία Ντάφνη Κόλτερα από ένα Αμερικανικό Πανεπιστήμιο και πραγματικά Είδα οι δυνατότητες που υπάρχουν στα Αμερικανικά πανεπιστήμια όσον αφορά την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος ή μίας διάλεξης μπορούν να παρακολουθήσουν ακόμα και χίλιοι φοιτητέ από όλες τις γωνιές του, του κόσμου. Και γνωρίζετε ότι πολλά Αμερικανικά πανεπιστήμια χρησιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο έχουν πετύχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Ας μην ξεχνάμε τα σημαντικότερα λοιπόν ωφέλη της εξαποστάσεως εκπαίδευσης, όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση σε όλο και περισσότερους φοιτητές. Δημιουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, μια παγκόσμια τάξη. Δεν χρειάζεται κανείς να ταξιδέψει μεγάλες αποστάσεις προκειμένου να παρακολουθήσει συγκεκριμένες διαλέξεις. Δεν χρειάζεται κανείς να κτίσει τεράστια πανεπιστήμια και αφιθέατρα προκειμένου να στεγαστούν όλοι αυτοί οι φοιτητές. Να σας δώσω κάποια ακόμα παραδείγματα. Ξέρετε ότι από το 1985 μέχρι σήμερα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ και οι τιμές των διδάκτρων και οι τιμές της κοινωνικής πρόνοιας και τα δίδακτρα τα ίδια έχουν αυξηθεί κατά, πολύ, κατά ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσοστό. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι η πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα από οικονομική πλευρά έχει μειωθεί για πάρα πολλού πολίτε. Μία λύση λοιπόν στο πρόβλημα αυτό των δαπανηρών ουσιαστικά σπουδών είναι η εξαποστάσεω εκπαίδευση. Ένα άλλο όφελο τη εξαποστάσεω εκπαίδευση και τη συμπληρωματική εκπαίδευση είναι η εξατομίκευση πλέον ορισμένων μαθημάτων. Ο φοιτητή δεν είναι πλέον απλώ ε, ένας αριθμός, η εκπαίδευση γίνεται όλο και πιο εξατομικευμένη και αυτό ισχύει και για τα εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία επιλέγουν οι φοιτητέ. Το ότι χρησιμοποιούνται επίση οι νέε τεχνολογίε πληροφορική αποτελεί εκ των ουκάνευ προπόθεση προκειμένου να μπορεί να ευοδοθεί αυτή η νέα μορφή εξ αποστάσεω εκπαίδευση. Η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων συσκευών και άλλων τεχνολογιών μα επιτρέπει να υποφεληθούμε πλήρω από τη νέα αυτή μέθοδο διδασκαλία. Και ένα ακόμα όφελο είναι η εκπαίδευση υψηλή ποιότητα που απορρέει από τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα. Θεωρώ ότι οι φοιτητέ κατά αυτόν τον τρόπο συμμετέχουν πολύ περισσότερο οι ίδιοι στα εκπαιδευτικά προγράμματα, με αποτέλεσμα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται όλο και πιο ποιοτικό. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το εκπαιδευτικό μοντέλο είναι όλο και πιο πολλά υποσχόμενο, σε σημείο που θα μπορούσαμε για κάποιους τομείς να εγκαταλείψουμε ακόμα και τα παραδοσιακά μοντέλα εκπαίδευσης. Θεωρώ ότι μπορούμε χρησιμοποιώντας τις νέες αυτές μεθόδους να προσδώσουμε νέες γνώσεις και νέες δεξιότητες σε όλο και περισσότερους πολίτες. Προσβλέπω στη σύνταξη λοιπόν της έκθεσης αυτής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις σημαντικές σας παρατηρήσεις και εν κατακλείδη θα ήθελα να αφαιρθώ σε δύο σημαντικότατα ζητήματα που κατά την άποψή μου είναι πρωτοφανή και απορρέουν και από αυτά που μας είπατε. Η διαβίου μάθηση είναι ουσιαστικά το, η πίστη που έχουμε στην ε, όλο και μεταβαλλόμενη αυτή κοινωνία πρέπει να μπορούμε ήδη από τώρα να προβλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε τις νέες αυτές εξελίξεις που θα έχουμε στο μέλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι πολίτες να έχουν όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση στην άτυπη και μη τυπική μάθηση, παράλληλα με την κλασική παραδοσιακή εκπαίδευση. Αυτές οι νέες μορφές εκπαίδευσης, συμπληρωματική και εξ πραγματικά είναι δύο μορφές πολλά υποσχόμενες για όλους τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις σας και το παραλαμβάνω για μία ακόμα φορά. Είναι ιδιαίτερα πολύτεμες και θα συμβάλλουν πάρα πολύ στην κατάρτιση της έκθεσής μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σβέρ, πρώτα θα ακούσουμε τώρα τους και ηγητές, στο βαθμό που είναι παρόντες βέβαια, και μετά άλλους τους υπολείπους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Θα πρότεινα χρόνο αγόρευσης 3-4 λεπτά. Αν στο τέλος έχουμε χρόνο, δεν θα κάνουμε και ένα δεύτερο γύρο τοποθετήσεων. Έτσι να γίνει πιο πολύ συζήτηση. Ο κύριος Νέκοφ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τα τελευταία δυόμιση χρόνια ήρθε σε επαφή με πάρα πολλούς νέους και είδα ότι αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, σε χώρες σαν τη δικιά μου, τη Βουλγαρία. Και ένα βασικό τους πρόβλημα είναι ουσιαστικά η διαρροή εγκεφάλων. Πάρα πολλοί νέοι αυτή τη στιγμή ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους, πάνε και εργάζονται σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Συνεπώς πιστεύω ότι μέσω των νέων τεχνολογιών μπορούμε να παρέχουμε εξ αποστάσεως εκπαίδευση στους ανθρώπους αυτούς προκειμένου να μπορούν να εργάζονται και παράλληλα να εκπαιδεύονται περαιτέρω, να κερδίζουν όλο και περισσότερες δεξιότητες και γνώσεις από τα πανεπιστήμια της Δυτικής Ευρώπης, να μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα ανταλλαγής, να συμμετέχουν σε κοινέ διαδικτυακές πλατφόρμες εκμάθησης, πλατφόρμες του 21ου αιώνα που φέρνουν από κοινού πολλές διαφορετικές ιδέες και πολλά διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό που μας είπε ο κύριος Χόιερ είναι ειδικά πολύ σημαντικό. Οι συστάσεις στις οποίες προχώρησε είναι πολύ σημαντικές και πολύ σημαντικές είναι οι συστάσεις του κυρίου Ούμπαξ επίσης. Μπορούμε κατά αυτόν τον τρόπο να δίνουμε στους νέους νέες επιλογές, νέες εναλλακτικές εκμάθησης και περαιτέρω κατάρτισης. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις νέες τεχνολογίες προκειμένου να γνωρίσουμε και νέες μορφές διδασκαλίας όντας σε επαφή και με τα πανεπιστήμια αλλά και με την επιχειρηματική κοινότητα. Πριν από ορισμένου μήνε έγινε και μία δημόσια ακρόαση. Νομίζω στην Τοσκάνη. και μάθαμε εκεί πέρα ότι στην περιφέρεια αυτή της Ιταλίας υπήρξαν πάρα πολλές start-up επιχειρήσεις οι οποίες επωφελήθηκαν από τα διαδικτυακά προγράμματα εκμάθησης τα οποία προωθούσαν τα πανεπιστήμια της περιοχής. Νομίζω λοιπόν ότι συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συνεργασία με τις ίδιες επιχειρήσεις, όλο και περισσότεροι νέοι θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες, σε νέα προγράμματα κατάρτισης και εκμάθησης. Και να πω και κάτι ακόμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από τη χώρα μου, τη Βουλγαρία. Τα περισσότερα πανεπιστήμια στη χώρα μου βρίσκονται στη Σόφια, στην πρωτεύουσά μας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Όταν αποφυτεί κάποιος από το Πανεπιστήμιο της Σόφιας, για παράδειγμα, κατά πάσα πιθανότητα ο απόφυτος αυτός θα παραμείνει στην πρωτεύουσα και δεν πρόκειται να επιστρέψει στην ιδιαίτερη πατρίδα του. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Χέλγα Τρούπελ. Ευχαριστώ, ε, Να ευχαριστήσω και τους προσκεκλημένους μας που ήταν πολύ ενδιαφέρον τους ακούσαμε. Είδαμε τι δυνατότητες μας ανοίγει η ψηφιοποίηση, το άνοιγμα των πανεπιστημίων, ώστε να μπορούν να προσαγγίσουν πολύ μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού. Μιλούμε για την κοινωνία της γνώσης και είναι σαφές ότι το δυναμικό των πανεπιστημιακών φορέων εδώ δεν μπορούμε να θεωρούμε ότι έχει εξαντληθεί για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι μας καλείται αυτές τις δυνατότητες να τις συμπεριλάβουμε και να τις ενσωματώσουμε στις ε, δυνατότητες προεπολογισμού χρηματοδότησης που έχουμε, ώστε να δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες σε τέτοιες προσεγγίσεις. Και επίσης, κάτι που δεν είναι καινούριο για εμάς, αλλά είναι σημαντικό να το επαναλάβουμε, ότι πρέπει να έχουμε μια ισότιμη αντιμετώπιση στην αναγνώριση των επίσημων μορφών εκπαίδευσης και των άτυπων μορφών. Σχετικά λοιπόν με αυτήν την ε, επαφή με τους νέους και με μεγαλύτερες ομάδες του πληθυσμού, αυτό που δεν μου είναι απόλυτα σαφές είναι τι έχετε κάνει με στιγμής, αν έχετε κάνει κάτι, αν έχετε κάποια μεγέθη σχετικά με την ισότητα των φύλων. Πώς αυτό δηλαδή έχει αποτυπωθεί στους διαφόρους τομείς της δουλειά που έχετε κάνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χέλγα. Η κυρία Κώστα. Νομίζω ότι σήμερα το απόγευμα ε, είχαμε υψηλότερο ενδιαφέρον χάρη στις εισηγήσεις σας, ε, οι οποίες ε, συμπλήρωναν η μία την άλλη και μας έδιναν ένα πλήρες πλαίσιο αφιερωθήκαμε σε μια γνωμοδότηση πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου γιατί είναι όριμη η στιγμή και όπως μας συστήνεται και εμείς πρέπει να διατηρήσουμε ένα πλαίσιο για να αναπτύξουμε και ένα νοηματικό ακόμα πλαίσιο της στρατηγικής ψηφιοποίησης του θεματολογίου των δεξιοτήτων και της επερχόμενης ανακοίνωσης τη για τον εξυγχρονισμό της ανώτης εκπαίδευσης. Νομίζω ότι το θέμα εντάσσεται σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο τρία ερωτήματα που ήθελα να σας θέσω. Σχεδόν όλοι και να ευχαριστήσω για τη διάκριση στον παρόδο μεταξύ του τι είναι μέθοδος και τι είναι περιεχόμενο κάποιων μορφών εξ αποστάσεως ε, εκπαίδευσης ως συμπληρωματική μορφή εκπαίδευσης. Ε, ένα πρώτο ερώτημα λοιπόν. Εμείς έχουμε τρόπον ένα πλαίσιο αναγνώρισης Τη επίσημη, ανεπίσημη και άτυπη εκπαίδευση. Εσεί θεωρείτε ότι αυτό δίνει ανεπαρκέ ανεπαρκές απέναντι σε διάφορα πρότυπα που επιτρέπει η εξαποστάσεω φίτηση σήμερα. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών, των κρατικών φορέων διασφάλισης ποιότητας κτλ. Μας προτείνεται λοιπόν να υπάρχει ένα πιο συγκεκριμένο πλαίσιο απέναντι στην ασφάλεια που είναι σημαντικό σημείο, την προστασία των δεδομένων, αλλά και της αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων. Επομένως, είναι σημαντικό να καταλάβουμε ποια είναι τα συγκεκριμένα βήματα που πρέπει να αναλάβουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ε, το δεύτερο ερώτημα αφορά στη δυνατότητα αναγνώρισης μεταξύ μάλλον. Εσείς μιλάτε για εξαποστάσεως εκπαίδευση ως συμπληρωματικό πρόγραμμα. Υπάρχουν στη χώρα μας και νομίζω και σε άλλες χώρες, έχουμε και τον σύλλογο που εκπροσωπείται εδώ, ε, ε, προγράμματα ε, αποκλειστικά εξαποστάσεως φίτησης. Επομένως, η ερώτηση είναι μεταξύ του Open University ή άλλων φορέων πανεπιστημίων που παρέχουν τέτοια προγράμματα, η δική σας αρμοδιότητα ή εμπειρογνωμοσύνη είναι να μεταφέρετε αυτήν την γνώση και σε πανεπιστημιακούς φορείς που ενδεχομένως να μην έχουν προσανατολιστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Και μιλά, αναφέρομαι και στο τελευταίο συνέδριο που είχαμε ε, το Νοέμβριο στη Ρώμη σχετικά με την εμπειρογνωμοσύνη των πανεπιστημίων, των κάμπους, των πανεπιστημιακών χώρων που έχουν ένα έλλειμμα ενδεχομένως τέτοιων προγραμμάτων. Και τελευταίο, το θέμα των σπουδαστών και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και η μελέτη που κάνατε και από ό,τι κατάλαβα καλά, εμείς θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε τέτοια προγράμματα και για τους ενήλικες ή για στοχευμένες ομάδες πληθυσμού. Επομένως η αναγνώριση αυτών των ε, ε, σύντομων προγραμμάτων σπουδών ε, έχω την εντύπωση ότι είναι ένα από τα ζητήματα κλειδιά. Και σε αυτό το επίπεδο ποιο θα μπορούσε να είναι το ευρωπαϊκό πρότυπο είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σότροβα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχά θέλω να σας ευχαριστήσω. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι παρουσιάσεις και θα βασίσουμε την επόμενη εργασία μας ε, σε αυτά που ακούσαμε. Πραγματικά σας ευχαριστώ όλους. Μερικά σχόλια έχω και ερωτήσεις να κάνω. Αυτό που είπατε κύριε Χόιερ για τους δασκάλους που θα πρέπει να γνωρίζουν ε, από επικοινωνία και μίντια. Αυτό είναι πολύ βασικό αν θέλουμε να προετοιμάσουμε τους αυριανούς πτυχιούχους ε, δευτεροβάθμιας και τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει η εξαποστάσεως εκπαίδευση και διδασκαλία, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει οι δάσκαλοι να έχουν τα προσόντα και τις δεξιότητες, άρα υπάρχει πρόσβαση σε αυτά και να υπάρχει και το σωστό ακαδημαϊκό πλαίσιο και, και μαθησιακό και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους ακαδημαϊκούς δασκάλους, αλλά και για τους καθηγητές ε, της δευτεροβάθμιας και τους δασκάλους πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Και θέλω να ρωτήσω και την κυρία Κλίνκνερ, η οποία μας έθεσε πέντε στόχους και πέντε ε, αιτήματα. ότι θα πρέπει να αναγνωρίζεται η συνέχεια και η διαρκής εκπαίδευση ε, ως βασικός ρόλος του Πανεπιστημίου με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Μα ξέρετε ότι τα πανεπιστήμια είναι αυτόνομα σε πολύ μεγάλο βαθμό και έχουν και ε, δική τους δομή και διοίκηση. Το συζητούν μεταξύ τους τα πανεπιστήμια. Η δική σας ε, οργάνωση ή απλώς καταλήξατε σε αυτό το συμπέρασμα μετά από έρευνα. Έχουν κάποια αυτοτέλεια τα πανεπιστήμια. Ε, και το ε, Erasmus, ε, το Erasmus Plus είναι καλό να χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και για την εξαποστάσεως εκπαίδευση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Σόπφλιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστίες προς όλους τους προσκεκλημένους σας με τα πολύ ενδιαφέρουσα που μας είπαν. Εγώ μία τριακονταετία πέρασα στην ανώτερη εκπαίδευση, στα υψηλότερα κλιμάκια ενδεχομένως. Και έχω τρία ερωτήματα. Το πρώτο είναι προς τον καθηγητή Χόια, ίσως να διαφωνήσει μαζί μου. Κατά τη δική μου εμπειρία, περί το 95% των σπουδαστών σπουδάζουν προκειμένου να αποκτήσουν ένα τίτλο, ένα δίπλωμα, ένα πτυχίο. Αυτό που λείπει είναι η επιστημονική περιέργεια που κινεί έναν ακαδημαϊκό να συνεχίσει να ψάχνει, να ερευνά. Και κατά πόσον βοηθάει σε αυτό η ψηφιοποίηση. Υπάρχει λοιπόν μια χαρτογράφηση αυτής της πνευματικής περιέργειας, της ακαδημαϊκής περιέργειας, και ήθελα να καταλάβω κατά πόσον συνδέεται αυτό με την ψηφιοποίηση. Προς τον κύριο Hetherington ε, αναφέρατε ένα 11% εθνικών μειονοτήτων ενδεχομένως ε, συμπεριλαμβάνεται τις εθνικότητες στην Ευρώπη. Ούγγρους, Πολωνούς, Ρουμάνους και τα λοιπά και τα ποσοστά τους σε άλλες χώρες. Επίσης, τα ποσοστά που αναφέρατε σχετικά με τον αλφαβητισμό ε, ποια είναι τα κριτήρια επιτυχίας εκεί. Πώς γνωρίζετε ότι έχετε επιτύχει τα επίπεδα του αλφαβητισμού που απαιτούνται είτε από τη δική σας οπτική σκοπιά είτε του CPI. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σοφλή. Η Κριστίνα Λιμπάτσκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όντως, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους εμπειρογνώμονές μας για τις πολύ ενδιαφέρουσες αυτές παρουσιάσεις. Είναι διτές, θεωρώ, οι ερωτήσεις που τίθενται αυτή τη στιγμή. Καταρχά, το επίπεδο γνώση που έχει κανεί και το πόσο εύκολα απαρχαιώνεται το επίπεδο γνώσης που έχει, το πτυχίο ενδεχομένω στο δίπλωμα και πώ μπορούμε να συμπληρώσουμε λοιπόν τι δεξιότητε και τι γνώσει μα προϊόντο του χρόνου. Οι νέε πληροφορίε επίση είναι πολύ εύκολα προσβάσιμε. σας μην το ξεχνάμε αυτό και σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριο Χόιερ. Είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξη όταν βλέπω να αναδύονται νέε ευκαιρίε. όταν έχουμε νέε μορφέ πανεπιστημίων όπω το ανοιχτό πανεπιστήμιο, νέες μορφές εκμάθησης και εκπαίδευσης. Δεν θα ήθελα όμως το Πανεπιστήμιο του Μέλλοντος να αποτελεί ένα Πανεπιστήμιο Google, όπως είπε ο καθηγητής Χόιερ πριν από λίγο. Α μην χαθεί λοιπόν και το παραδοσιακό πανεπιστήμιο. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε ένα πραγματικό πανεπιστήμιο και το πανεπιστήμιο Google. Το πανεπιστήμιο Google προσφέρει απλώ πληροφορίε. Το κλασικό παραδοσιακό πανεπιστήμιο προσφέρει γνώση, ουσιαστική γνώση. Νομίζω λοιπόν, με όλο το σεβασμό που έχω βέβαια για τις απόψει σας και για τις νέε μορφές πανεπιστημίων, αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και καθοριστική σημασία είναι η ποιότητα. Πολύ καλή πρόσβαση σε πληροφορίες, αλλά μην γίνεται αυτό ει βάρος της παρεχόμενη παιδεία και της ποιότητας παρεχόμενη παιδεία. Ένα οποιοδήποτε πιστοποιητικό μπορεί να παρέχεται, επίσημη ή ανεπίσημα, αλλά είναι ανυπόστατο το πιστοποιητικό αυτό αν πραγματικά δεν βρίσκεται από πίσω το ένα υψηλό επίπεδο ουσιαστική γνώση. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να μα απασχολήσει και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προστατεύσουμε και τι παραδοσιακέ πανεπιστημιακέ μορφέ. Και πέρα από αυτό, όσο περνάει ο χρόνο, θα πρέπει να εξασφαλίζουμε την ε, υψηλότατη παιδεία της κατάρτισης των ίδιων των διδασκόντων, των ίδιων των καθηγητών. Γιατί άλλο πράγμα να πρέπει να αποκτά κανείς γνώση και άλλο πράγμα να πρέπει να διαβιβάσει και να μεταβιβάσει μάλλον κανείς, να μεταναμπαδεύσει τη γνώση και τις δεξιότητες. Ενδεχομένω να σα προκαλώ αυτή τη στιγμή κάπω με τι απόψει μου. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση και προ τον εισηγητή. Ενδεχομένω στην έκθεσή σα να μπορέσετε να φερθείτε στις ειδικέ ακαδημαϊκές ζώνες του ανοιχτού πανεπιστημίου και στις νέες προϋποθέσεις και τις απαιτήσει προκύπτουν. Η επαγγελματική κατάρτιση είναι ένα πράγμα, αλλά όταν εστιαζόμαστε στο ζήτημα αυτό, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι και η απόκτηση των δεξιοτήτων είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά θα πρέπει να εξισορροπείται με την ίδια τη γνώση η καλύτερη δυνατή ισορροπία μεταξύ γνώσης και δεξιοτήτων. Χωρίς γνώση δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να υποφεληθούμε από τις δεξιότητες που έχουμε αποκτήσει. Και τέλος, οποιαδήποτε έκθεση και αν έχουμε καταρτήσει, διαδικασία Μπολόνια, διάμεση αναθεώρηση για το πρόγραμμα Εράσμους, κάθε φορά σε όλες αυτές τις εκθέσεις να φερόμαστε στις νέες ευκαιρίες οι οποίες συνδυάζονται με τα νέα μέσα, με τα ανοιχτά πανεπιστήμια και το καθεξής. Αλλά πάντα, πάντα λέμε ότι ε, μπορούν σαφώς να αλλάξουν το χαρακτήρα της διαδικασίας στην Πολόνια όλες αυτές οι νέες μέθοδοι. Και πάλι αυτό μπορεί να γίνει όμως μόνο αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την κατάλληλη διεπαφή ανάμεσα στα δύο, δεξιότητες και γνώση. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να καταλήξουμε σε νέες διεπιστημονικές διαδικασίες, οι οποίες είναι πάρα πολύ, σημαντικές για την πρόθεση, πολύ σημαντικές για την πρόθεση της ίδιας επιστήμης. Και αυτό αποτελεί πρόκληση για όλα τα πανεπιστήμια. Πρέπει τα πανεπιστήμια που από τις νέες τεχνολογίες να είναι σε συνεχή επαφή το ένα με το άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ξεπεράσατε λίγο τα τέσσερα λεπτά, λίγο όμως, εντάξει, όλα καλά. Ε, θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλει να λάβει θέση. Gerne, Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Εκεί ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, ευχαριστήσω όλα τα μέλη του πάνελ για, πολύ, για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και εισηγήσεις τους. εγώ θα σας πω τι κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι σχεδιάζουμε. Αναφέρθηκε ήδη ότι αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε στην επικαιροποίηση του εξυγχρονισμού του θεματολογίου για την ανώτερη εκπαίδευση. Περιμένουμε αυτό να δημοσιευθεί προς τα τέλη Μαΐου. Στη δημόσια διαβούλευση έρευνα που κάναμε πέρυσι για την ψηφιοποίηση και την παγκοσμιοποίηση προέκυψε σαφώς ότι αυτά τα δύο στοιχεία είναι βασικοί παράγοντες πρόοδου σχετικά με την παροχή της ανώτητης εκπαίδευσης, ποιος την παρέχει, ποιος τη λαμβάνει, για την ποιότητα των καθηγητών επίσης και των προγραμμάτων ε, των εκπαιδευτικών και εδώ στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα συμπεριλαμβάνουμε όλα τα ιδρύματα που παρέχουν εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών η συνεισφορά τους στην καινοτομία και για να σας δώσω κάποια μεγέθη, το 45% των απαντήσεων εκφράζουν ανησυχίες ότι η τεχνολογία δεν, ε, δεν εφαρμόζεται, δεν χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και το 90% αναφέρεται στην ανάγκη του να επικαιροποιήσουμε, να αναπτύξουμε, το, μάλλον να βελτιώσουμε το επίπεδο του καθηγητικού προσωπικού έγινε μια διαβούλευση μεταξύ 15 κρατών μελών για το πώς η ψηφιοποίηση μεταβάλλει το τοπίο της μάθησης, της εκπαίδευσης. Για το Erasmus Plus και το πρόγραμμα εργασίας του 2017, το οποίο έχει συγκεκριμένες αναφορές στις ε, ψηφιακές δεξιότητες και στην παροχή στήριξης για έργα συνεργασίας μεταξύ της ανοιχτής εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Υπάρχει επίσης συγκεκριμένη μνήμα σε στήριξη για έργα που προσπαθούν να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την αναγνωρισιμότητα των ε, τίτλων σπουδών. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι ζήτημα. Σχετικά με τη διασφάλιση ποιότητας, Στι ερχόμενε εβδομάδες ε, θα ξεκινήσουμε έναν επόμενο διαγωνισμό για μια έκθεση πλαισίου που θα ενημερώνει, που θα τροφοδοτεί μάλλον την επόμενη έκθεση για την διασφάλιση ποιότητα ε, που η Κομισιόν θα υποβάλει σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Εκεί εξετάζουμε ιδιαίτερα ενδελεχώς την ψηφιοποίηση, όπως και τα πορίσματα του κομμουνικέ του 2015 που εξέδωσαν οι Υπουργοί για την διασφάλιση ποιότητα σύμφωνα με τις κατευθύνες γραμμέν με ιδιαίτερο στόχο να ανταποκριθούν σε μια υψηλή προσδοκία τα πανεπιστήμια, τα πανεπιστήμια να, γίνουν, να επικεντρωθούν περισσότερο στους σπουδαστέ, να επικεντρωθούν στους νέους, στις νέες μορφές ε, παράδοσης περιεχομένου δηλαδή τις ψηφιακές όλα αυτά όταν θα έχουν ολοκληρωθεί θα τροφοδοτήσουν ακριβώς την έκθεση που θα υποβάλουμε σε εσά όπως και στο Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, θα ήθελα να ξαναδώσω το λόγο στους ε, προσκεκλημένους εμπειρογνώμονες για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που ανέκυψαν ή να κάνουν και κάποια σχόλια ε, σε όσα άκουσαν από τους βουλευτές. Να αρχίσουμε με την αντίστροφη σειρά τώρα θα πρότεινα. Πρώτος ο κύριος Ούμπαχς. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάω λίγο τις ερωτήσεις αυτή στην οποία μπορώ να απαντήσω άμεσα είναι η ερώτηση της Σίλβια Κώστα. Πώς η εξαποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να έρθει να συμπληρώσει τα παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εμπειρία συσσωρευμένη από τα νέα πανεπιστήμια, τα καινοτόμα, για να βοηθηθούν τα κλασικά παραδοσιακά πανεπιστήμια. Το ερώτημα αυτό ετέθηκε προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από κάποια χρόνια σε σχέση με το θεματολόγιο εξυγχρονισμού. Επικεντρωνόμαστε αυτή τη στιγμή στη διδασκαλία, ιδίως στα πλαίσια των πανεπιστημίων εκείνων που παρέχουν προγράμματα διδασκαλίας εκμάθησης εξ Μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε στην έρευνα που έχει γίνει και στην πείρα που έχουν συσσωρεύσει τα πανεπιστήμια αυτά. Ξέρουμε ότι παράδειγμα το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Ηνωμένου Βασιλείου ή των κάτων χωρών έχουν συγκεκριμένα πλέον τμήματα για την καινοτομία στην εκπαίδευση. Και έχουν καταφέρει μέσω της έρευνας που έχουν κάνει στον τομέα αυτό και μέσω της εμπειρίας που έχουν συσσωρεύσει να διαμορφώσουν νέα εκπαιδευτικά μοντέλα, τα οποία έχουν διαβιβάσει και προς άλλα πιο κλασικά, αν θέλετε, πανεπιστήμια αλλού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Empowering Universities, ενίσχυση των πανεπιστημίων, όπου έχουμε εμπειρογνώμονες από διάφορα πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε 12 προγράμματα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συμπληρωματικών και εξαποστάσεως και έχουμε κατά αυτόν τον τρόπο, αν θέλετε, 12 διαφορετικές μορφές εμπειρογνωμοσύνης που έχουμε συγκεντρώσει με τη χρησιμοποίηση της ε, συμβολής διαφόρων πανεπιστημίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν, έχουμε διοργανώσει και σε τήσια βάση τρία webinars, σεμινάρια δηλαδή στο διαδίκτυο, τα οποία είναι ανοιχτά προς όλα τα πανεπιστήμια ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσπαθούμε ακριβώς να επικεντρωθούμε σε αυτές τις νέες μορφές, ε, τις μικτές μορφές διδασκαλίας, όπου καλούμε όλο και περισσότερους καθηγητές να ενημερωθούν για τα προγράμματα αυτά και να συμβάλλουν και οι ίδιοι. Κατά αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια γόνιμη ανταλλαγή ε, εμπειριών και γνώσεων και υπάρχουν και εμπειρογνώμονε οι οποίοι πηγαίνουν οι ίδιοι στα πανεπιστήμια εκείνα τα οποία δεν έχουν κάνει αυτή τη μετάβαση, το ποιοτικό αυτό άλμα προ τι νέε μορφέ διδασκαλία και εκμάθηση. Υπάρχει λοιπόν ένα ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο όπως σα είπα ονομάζεται Empowering Universities. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέχασα να το πω προηγουμένω. Δεν χρειάζεται να απαντάτε όλοι σε όλε τι ερωτήσει. Ψάξτε εκείνε που σα είχαν απευθύνει οι συνάδελφοι, ή θεωρείτε ότι μπορείτε να απαντήσετε και να συνεισφέρετε κάτι χρήσιμο. Η κυρία Κλίνκνερ. Yeah, yeah. Ναι. Καταρχάς, θα ήθελα να απαντήσω ε, σε αυτό που ρωτήσατε για το φύλλο, ε, για τους συμμετέχοντες, αν υπάρχει καμιά ιδιαίτερη κατανομή στην εξαποστάσεω σπίτι. Τώρα δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμηριωμένα, ε, μαζί μου, αλλά εμείς τη διαπιστώνουμε στο σύλλογό μας ότι ε, φτάνουμε καλύτερα στις γυναίκες ε, γιατί μπορούν να συνδυάσουν την οικογένεια και το επάγγελμά τους και τον εργασιακό τους βίο με τις σπουδέ από τη στο κλασικό πανεπιστήμιο. Ή στην πληροφορική ε, συμμετέχουν περισσότερες γυναίκες στην εξαποστάσεως εκπαίδευση από ό,τι στη φοιτηση στο πανεπιστήμιο, ακριβώς γιατί είναι πιο εύκολο να το κάνουν από το σπίτι τους κτλ. Άρα ταιριάζει και με τους στόχους που έχουμε βάλει για ευρύτερη διαφοροποίηση και εκπροσώπηση περισσότερων ομάδων ε, του πληθυσμού. Μεγάλο πλεονέκτημα και αυτό. Μετά, να απαντήσω σε μια ερώτηση που είχε να κάνει λίγο με διάφορα σημεία που προβάλλουμε εμείς ως αιτήματα από την οργάνωσή μας. Πώς μπορούμε αυτό να το συνδυάσουμε με την επιστημονική ελευθερία και την, το αυτοδίκητο πούμε, των πανεπιστημίων. Ε, είναι προφανές ότι ε, συνεννοούμαστε και για τις, με τις προδιαγραφές και με τα πανεπιστήμια και με τους διαφόρους εκπροσώπους. Δεν είναι τυχαία αυτά τα αιτήματα και ουρανοκατέβατα. Είναι η καθημερινότητά μας. Ε, αυτά μας τα θέτουν τα πανεπιστήμια. ότι και τα κλασικά παραδοσιακά πανεπιστήμια που ο ε, επιτόπου ε, προσφέρουν και εξ αποστάσεως τμήματα και προγράμματα σπουδών. Και στη δική μας οργάνωση εμείς υποστηρίζουμε 18 ε, πανεπιστήμια υποχρεωτικής φοιτής ας πούμε, αλλά που έχουν και εξ αποστάσεως προγράμματα και ο πρόεδρος του συλλόγου μας ηγείται ε, στη Ρινανία Παλαντινάτου σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα τέτοιο τμήμα εξ αποστάσεως. Δηλαδή, ε, μας απασχολούν ε, αυτά, δεν είναι ειδικά ξεχωριστά τα πανεπιστήμια εκείνα που προσφέρουν εξ αποστάσεως ε, εκπαίδευση και τίποτα άλλο. Υπάρχουν και τέτοια. Αλλά συνήθως τα κλασικά πανεπιστήμια ε, έχουν και τέτοια προγράμματα ε, σπουδών, αλλάζουν τα πράγματα και χαιρόμαστε γι' αυτό και βεβαίως συζητούμε με τα πανεπιστήμια αυτά, είμαστε σε επαφή και φροντίζουμε και διαπιστώνουμε άλλον ότι αλλάζουν και οι δομές στα κλασικά παραδοσιακά πανεπιστήμια όσο αλλάζουν τα πράγματα. Αυτά νομίζω αφορούσαν εμένα για να απαντήσω. Ευχαριστώ πολύ. Να πω και εγώ κάτι, έτσι ένα σχόλιο. Η ελευθερία της διδασκαλίας και της έρευνας και η διεύρυνση της νομοθετικής εντολής προς τα πανεπιστήμια και για τη διαβίου μάθηση να φροντίζουν δηλαδή, ε, δεν είναι ε, αντιφατικά, είναι συμπληρωματικά. Δηλαδή ε, το να ορίσει ο νομοθέτης ότι το πανεπιστήμιο έχει ένα ρόλο και διαβίου μάθηση, δεν σημαίνει ότι το περιορίζει στην ελευθερία τη διδασκαλία τη έρευνα και γενικά ε, του δένει στα χέρια. Ε, ο κύριο Χέδρικ τον έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να σχολιάσω σε πέντε ερωτήματα που ετέθησαν. Το ένα ήταν για την ισορροπία των φύλων. Το δεύτερο για το λεγόμενο πανεπιστήμιο Google ε, το τρίτο για κάποιες προκλήσεις για την ακαδημαϊκή ελευθερία και τέταρτο και πέμπτο τα δύο συγκεκριμένα που με ρώτησαν για την παρουσίασή μου. Ε, κοιτάξτε, η δική μας εμπειρία για την ισότητα των φύλων είναι αντίστοιχη με εκείνη που εξέφρασαν οι δύο προηγούμενες, προηγούμενοι ομιλητές. Υπάρχει πολύ μεγάλη απόκληση ανά αντικείμενο, ανά πρόγραμμα σπουδών και οπωσδήποτε εμείς αυτό που έχουμε βρει είναι ότι σε κάποια αντικείμενα και εδώ σκέφτομαι περισσότερο τις κοινωνικές σπουδέ, υπάρχουν σημαντικά περισσότερες γυναίκες παρά άνδρες στην κοινωνιολογία, στις εξειδικεύσεις που έχουν σχέση με τους νέους, σε άλλες κοινωνικές σπουδέ. φαίνονται όλα αυτά να είναι πολύ πιο ελκυστικά ως αντικείμενα στις γυναίκες. Εκεί που έχουμε τη βασική πρόκληση, και θα συμφωνούσα με τους προηγούμενους, είναι στις θετικές επιστήμες και στους μηχανικούς, όπου έχουμε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ανδρών. Όμως θα συμφωνούσα με το σχολείο των προηγουμένων ομιλητών ότι η εξαποστάσεως ε, σπουδή είναι πιο ελκυστική σε αυτά τα παιδεία για τις γυναίκες και πολύ συχνά είναι και πολύ πιο υποστηρικτική με άλλες οικογενειακές ευθύνες που πολύ συχνά έχουν οι γυναίκες μαζί με τι σπουδέ του. Και επομένω είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος να τις προσελκύσουμε σε αντικείμενα και πανεπιστημιακές σχολέ που παραδοσιακά ε, είναι λιγότερε από ότι οι άνδρες. Νομίζω ότι εκεί λοιπόν μπορεί η ω φίτηση να παίξει ένα ρόλο. Για τη διχοτομία τώρα ή την αντιπαράθεση αυτή, την ανάλυση μεταξύ ανοιχτού πανεπιστημίου, πανεπιστημίου Google κτλ. Θα μπορούσα εδώ να υποθέσω απλώς το εξής. Εκεί όπου έχουμε δει οποιασδήποτε ψηφιακές παρεκκλήσεις με την Apple, με το Uber, με οποιαδήποτε μεγάλη εταιρεία που έχει παρέμβει επιθετικά σε έναν τομέα. Ε, η τυπική περίπτωση είναι μια πλατφόρμα, ένας πάροχος πλατφόρμα, δηλαδή στην οποία μπορεί να προσέλθει οποιοδήποτε να συνδεθεί ένας πάροχος, αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο σε ένα τομέα. Η Amazon είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατηγορίας. Θα περίμενα λοιπόν ότι αυτό που θα δούμε όλο και περισσότερο στην εκπαίδευση στην επόμενη δεκαετία είναι μια επέκταση δομών πλατφόρμας όπου μπορεί να φιλοξενείται περιεχόμενο, να πιστοποιείται από φορείς που έχουν πανεπιστημιακή ε, αδειοδότηση και από παρόχους που μπορούν να λάβουν αυτό το περιεχόμενο και με την κατάλληλη πιστοποίηση να το παρέχουν μέσω μιας δομής πλατφόρμας. Εκεί θα έχουμε πολλά προβλήματα. Θα έχουμε προβλήματα αναγνώρισης, ε, προβλήματα ε, διασφάλισης ποιότητας και θα είναι πιθανότατα μια πολύ επιθετική παρουσία, εμφάνιση, εισαγωγή στον τομέα της ανώτητης εκπαίδευσης. Και αυτό το βλέπουμε ήδη σε κάποιες μορφές άτυπης γνώσης. Ε, έχουμε ήδη μια πλατφόρμα που λέγεται Future Learn, που, στην οποία συμμετέχουν 90 πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που παρέχουν δωρεάν ε, πόρους ανοιχτών προγραμμάτων μάθησης. Ακόμα αυτά δεν έχουν πιστοποιηθεί, είναι άτυπα, αλλά βλέπουμε συγκεκριμένες κινήσεις προς την κατεύθυνση της αναγνωρισμένης εκπαίδευσης. Και σχετικά με την ακαδημαϊκή ελευθερία, Υπάρχει ένα πολύ ευρύ φάσμα πραγμάτων που μπορεί να πει κανείς. Ε, το καθεστώς της αυτονομίας του πανεπιστημίου, ε, μια χάρτα ενδεχομένως, ε, μια σημαντική πρόκληση εδώ και που και εσείς μπορείτε να έχετε σημαντική επιρροή να ασκήσετε στους πανεπιστημιακούς φορούς, φορείς είναι αυτή που σχετίζεται με το με τις αυτό που ονομάζουμε σήμερα αναγνώριση προηγουμένων σπουδών. Δηλαδή να ξεκινήσει ένας σπουδαστής σε μία πανεπιστημιακή σχολή, παραδοσιακή, στο χώρο του πανεπιστημίου, να εξασφαλίσει κάποιες ε, μαθησιακές πιστώσεις και να τις μετακινήσει σε ένα άλλο πανεπιστημιακό ίδρυμα ή άλλη σχολή και να συνεχίσει με διαφορετική κατεύθυνση. Υπάρχει όμως μεγάλος δισταγμός μεταξύ των πανεπιστημιακών φορέων ίσης αναγνώρισης των μαθησιακών αυτών πιστώσεων. Υπάρχει μια αντίσταση, αν θέλετε, ακαδημαϊκή σχετικά με την αναγνώριση των προηγουμένων σπουδών. Αυτό δεν είναι προς το όφελος των σπουδαστών. Και εδώ η διαβάθμιση ποιότητας είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά εμείς οπωσδήποτε θα ήμασταν υπέρ μιας προδραστικής προσέγγισης για να αναπτυχθεί η αναγνώριση των προηγουμένων σπουδών ή της προηγούμενης εγνώσης άλλης μορφής μη Τώρα σχετικά με τις ε, εθνικές μειονότητες, ε, αυτό που ρωτήσατε, δεν είμαι βέβαιος ότι ρωτούμε τόσο συγκεκριμένες πληροφορίες για την προέλευση κάποιου. Ε, χρησιμοποιούμε ένα ερωτηματολόγιο ώστε να ταυτοποιήσουν οι σπουδατές, οι σπουδαστές από πού είναι και μετά χρησιμοποιούμε διαφορετικά τα δεδομένα σχετικά με, την, ε, με τον κατάλογο των δεξιοτήτων CBI και πώς αυτό το χρησιμοποιούμε στα σπουδαστικά προγράμματα. Αυτό σχετίζεται με δύο μηχανισμούς. Πρώτον, ε, όλα τα πρότυπα σχετίζονται με ε, αν θέλετε πορίσματα γνωστικά, σπουδαστικά, παραδοτέα ώστε τελικά να επιτυγχάνεται ένα συνολικό αποτέλεσμα. Όταν τα καθορίζουμε αυτά τα πορίσματα, αυτά τα αποτελέσματα, τα κατηγοριοποιούμε με διαφορετικό τρόπο. Μερικά είναι συγκεκριμένα εστιασμένα ως προς το γνωστικό αντικείμενο. Και ως σπουδαστή πρέπει κανείς να μπορέσει να ε, επιδείξει, να αποδείξει τις γνώσεις του στη χημεία, στη γεωγραφία, στο δίκαιο, στο... σε οτιδήποτε είναι το αντικείμενο αλλά θα μπορεί κανείς από εκεί και πέρα και επί συγκεκριμένων τεχνικών, αν θέλετε, να δείξει τις επιδόσεις του, να δείξει τη σωρευμένη γνώση του ένας φοβαστής. Για παράδειγμα, κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε εξετάζοντας ας πούμε τις δεξιότητες επικοινωνίας, τα προσόντα τα επικοινωνιακά που είναι όλο και πιο σημαντικά για να είμαστε αποτελεσματικοί στον χώρο της εργασίας ίσως να είχαμε μια κοινή ανάθεση, ένα κοινό μάθημα σε μια ομάδα φοιτητών. Ε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να το εξετάσει κανός και ε, το δεύτερο που έχουμε εκεί είναι ένα πλαίσιο επιπέδων όπως το ονομάζουμε. Δηλαδή, στην όλη μαθησιακή ή σπουδαστική πορεία έχουμε διάφορα επίπεδα στην ε, ανάπτυξη των προσόντων με μια κίνηση προς ε, πιο ανεξάρτητη δυνατότητα σόρευσης γνώσεως. Προσπαθούμε λοιπόν να το συντροφεύσουμε στην πορεία αυτή όπου στο τέλος θα είχαν την δυνατότητα ε, ανεξάρτητα να δρουν. Ε, Βεβαίω, μια πτυχιακή εργασία, μια διπλωματική εργασία είναι το κλασικό, ο κλασικός τρόπος τον οποίο αποδεικνύει ένας σπουδαστή ότι έχει αναπτύξει αυτή την ικανότητα. Αλλά από εκεί πέρα υπάρχει και αυτή η γνωστική χαρτογράφηση στην οποία αναφερθήκατε που και αυτή χρησιμοποιείται προκειμένου να το καταδείξει αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταίος ο κ. Χόιερ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για το θέμα των πανεπιστημίων εξ αποστάσεως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα πανεπιστήμια αυτά να αναγνωρίζονται ως ισότιμα πανεπιστήμια με τα πανεπιστήμια που φυτά κανείς επιτόπου, από το κράτος δηλαδή, ότι έχουν τις ίδιες ε, προδιαγραφές, τα ίδια στάνταρ και τους ίδιους μηχανισμούς πιστοποίησης. Εγώ ε, δεν θεωρώ ότι το εξαποστάσεως πανεπιστήμιο είναι το πανεπιστήμιο της δεύτερης ευκαιρίας, γιατί δεύτερη ευκαιρία σημαίνει και δεύτερη ε, κατηγορία. Για πολλούς είναι η πρώτη ευκαιρία και η μοναδική ευκαιρία που έχουν να φτάσουν σε μια ακαδημαϊκή ζωή. Είναι πολύ σημαντικό η αποδοχή σε σχέση με τα φύλλα. 19 χρόνια ήμουν ε, στο Χάγκεν ε, Πρίτανης του ε, πανεπιστημίου εξ που με αριθμό φοιτητών είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στη Γερμανία και σε όλα ε, τα γνωστικά αντικείμενα είναι περισσότερες οι γυναίκες. Γιατί είναι γυναίκες που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους και θέλουν να ανακτήσουν τα προσόντα τους ή να αποκτήσουν νέα προσόντα για την αγορά εργασίας. Και ποια είναι η εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Εμείς θέλουμε οι φοιτητέ μας να βρουν δουλειά στην αγορά εργασίας. Αυτό είναι το κριτήριο και να έχουν μια ευκαιρία ανεξαρτήτως εκπαίδευσης και δρόμου που θα τους φέρει εκεί. Αναφέρθηκε το θέμα της προστασίας και της ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Βεβαίως πρέπει να το εξασφαλίσουμε. Υπάρχουν ε, τεχνολογικές ε, εξελίξεις ε, για την διδασκαλία και την εκμάθηση, learning analytics, για μια διάδραση ε, αλλά πολλές φορές προσκρούμε σε θέματα προστασίας δεδομένων και ε, πρέπει να το δούμε. Έγινε μια ερώτηση για το κατά πόσο τα εξαποστάσεως ε, πανεπιστήμιων μπορούν να δώσουν στα κλασικά πανεπιστήμια ιδέες για να προσαρμοστούν ε, στη σημερινή πραγματικότητα και στα δεδομένα. Αυτό μπορεί να γίνει μόνο επίσης όρης. Γιατί τα κλασικά έτσι, παραδοσιακά πανεπιστήμια δεν πρόκειται ποτέ να δεχτούν να έρθει ένα ε, επιγραμμικό να του πει τι να κάνουν. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ένα κάμπους, μια πανεπιστημιούπολη, μια πολυτεχνιούπολη ε, που υπάρχει τώρα στη Βόρεια Νέα που συνεργάζονται αυτά τα δύο είδη πανεπιστημίων. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι οι δεξιότητες ως προς την πληροφορική και τα μίντια των διδασκόντων. Αυτό θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ και στην επαγγελματική κατάρτιση και στον πανεπιστημιακό κόσμο να αξιοποιηθεί όσο γίνεται και να εξαντληθεί το δυναμικό της ψηφιοποίησης. Erasmus Plus το ανέφερε η Τζούλη ε, Άντερσον. Θα πρέπει να φροντίσουμε να καταλάβουμε το εξής. Όλο και περισσότερος κόσμος απελευθερώνεται από τους περιορισμούς που έχει, από την εργασία, από την οικογένεια και μπορεί να αποφασίσει να σπουδάσει εξ αποστάσεως. Δεν προσφέρεται το Erasmus Plus, γιατί χρειαζόμαστε κάτι που να διαρκεί τέσσερις εβδομάδες και όχι τέσσερις μήνες. Ο εργαζόμενος δεν θα αφήσει τη δουλειά του να πάει να κάνει ένα εξάμεινο σε ένα άλλο πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Και πού θα την ξαναβρει μετά. Δεν έχουν την πολυτέλεια να φύγουν από τη δουλειά τους έξι μήνες. Σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε εσεί κύριε Σόφλιν, είπα στην αρχή ότι ο ένας στους δύο από εμά θα τελειώσει τον επαγγελματικό του βίο σε άλλο επάγγελμα ε, από εκείνο που έχει αρχίσει. Όσοι αλλάζουν δουλειά ε, ε, θέλουν να πλατιάσουν, να βρουν ένα ε, άλλο στήριγμα να σταθούν, να μάθουν κάτι καινούριο. Όσοι μένουν στην ίδια δουλειά θέλουν να εμβαθύνουν, γιατί αυτά που έχουν μάθει στο πανεπιστήμιο πολύ γρήγορα είναι απαρχιωμένα. Εγώ αυτά που σπούδασα πριν από 35 χρόνια και 30 σήμερα ε, δεν θα μπορούσα να τα χρησιμοποιήσω, είναι τελείως άχρηστα. Δηλαδή αυτή η περιέργεια δεν χρειάζεται απλώς να ξυπνάει, να γεννιέται, αλλά να διατηρείται. Εξού και η ψηφιοποίηση που μας δίνει περισσότερες δυνατότητες από ό,τι στο παρελθόν που ήταν ε, ε, χρονικά περιορισμένη η διάρκεια της εκμάθησης, σπούδαζες, τελείωσες σπουδέ σου δούλευε. Και πάλι για τα πανεπιστήμια. Ε, στο μέλλον, κατά την άποψή μου, τι θα έχουμε. Οι προσφορές από εταιρείε για την αγορά εργασίας θα είναι πάρα πολύ ελκυστικές. Ο κόσμος δεν θα παίρνει πτυχίο από πανεπιστήμιο, αλλά πιστοποιητικό δίπλωμα από μια εταιρεία. Και θα πάνε μετά στο πανεπιστήμιο και θα πούνε αυτό πώς το βλέπεις, το αναγνωρίζεις που έχω από την εταιρεία. Εκεί παίζει αποφασιστικό ρόλο η ποιότητα. Αλλά θα πρέπει από τώρα να προετοιμαστούμε ότι είμαστε σε καιρούς παγκοσμιοποίηση και σιγά σιγά αυτά αναπτύσσονται και υπάρχουν και αιτήματα και αξιώσεις που θα γύρουν ορισμένοι στα πανεπιστήμια. Θα πρέπει τα πανεπιστήμια να το καταλάβουν και να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται σε αυτές τις νέες προκλήσεις. Αυτά και σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σφέρ, τον εισηγητή μας, αν θέλει να πει κάτι για να κλείσει ή όχι. Και εκείνος θα έχει τον τελευταίο, όχι για τον οριστικό, αλλά για σήμερα τον τελευταίο λόγο στον εισηγητή. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ που μου ξαναδίνετε το λόγο. Θα ήθελα να συνεχίσω στο σημείο που προλύσα σταμάτησε. Είπε ότι το παραδοσιακό κλασικό πανεπιστήμιο χάνει τη μονοπωλιακή του θέση πλέον σε αυτή τη νέα κοινωνία που βασίζεται στη γνώση και προκύπτουν τα νέα αυτά πανεπιστήμια τα οποία συντοποιούν όλο και περισσότερο ότι υπάρχουν νέες μορφές εκπαίδευσης οι οποίες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο. Θυμάμαι πριν από 10 χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ήδη από τότε να επεξεργάζεται κοινού ευρωπαϊκού μηχανισμού. Για παράδειγμα, ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων, αναγνώριση credits πανεπιστημιακών, αναγνώριση επαγγελματικών δεξιοτήτων, αναγνώριση προγραμμάτων επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Εγώ θυμάμαι ότι η Σλοβενία είχε υπογράψει ένα από τα προγράμματα αυτά όταν είχαμε τότε την Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την Προεδρία του Συμβουλίου. Ήταν τότε το πλαίσιο αναγνώριση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων κατάρτιση, επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ξεκινήσαμε την εργασία αυτή πριν από τόσα χρόνια. Θα πρέπει να τη συνεχίσουμε τώρα, ευθυγραμμίζοντα και να εναρμονίζοντα τι πρακτικέ μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντα ένα ενιαίο πλέον πλαίσιο όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτιση και εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά αυτό το οποίο βλέπω τελευταία χρόνια χάσαμε τον αρχικό μα αυτό δυναμικό ρυθμό δεν καταφέραμε να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση στην ανώτερη εκπαίδευση όσο θα έπρεπε. Και αυτό πραγματικά με στεναχωρεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πραγματικά γόνιμη η συζήτηση αυτή. Μας διαφώτισε πάρα πολύ, ιδιαίτερα για τη διαβίου Και μάθαμε πάρα πολλά Ήταν πάρα πολύ καλή ακρόαση, εξαιρετική και χάρη στους τέσσερις εμπειρογνώμονες που είχαμε προσκαλέσει που ο καθένας εξέτασε το θέμα από τη δική του σκοπιά και το φώτισε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Μας βοηθάει πάρα πολύ η παρουσία σας και η παρουσίασή σας. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. για τις ερωτήσεις, για τις παρατηρήσεις που μας βοηθούν να προχωρούμε πάντα. Και πριν ε, φύγετε όλοι και σχολάστε, να σας πω ότι η επόμενη συνεδρίαση είναι στις 27 Φεβρουαρίου, 3 με 6.30 και την άλλη μέρα με ψηφοφορίες 9 με 12.30. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το σημερινό απόγευμα και την υπόλοιπη συνεδρίαση και φυσικά και πάλι ε, ευχαριστώ τους ε, πυρογνώμονές μας και καλή επιστροφή ε, στα σπίτια σας. Ευχαριστώ και τις μεταφράστριες.